Καλημέρα σα, κύριε και κύριοι. Προσδεθείτε, ε, όχι, λάθο δεν πειράζει. Σας χαιρετώ όλους. Χαίρομαι που είσαστε τόσο πολύ πλησί σήμερα το πρωί και θα προσπαθήσω να αρχίσω σύντομα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ο εισηγητή δεν έχει έρθει ακόμα. Ελπίζω να έρθει σύντομα, γιατί έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος θα μας παρουσιάσει κάτι. Και καλωσορίζω την κυρία Ουξάντα Ντράγκλα Άγκλη. Άκλη, ελπίζω να είπα καλά το όνομά τη, η οποία είναι διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και χαίρομαι που είσαστε εδώ και μάλιστα στην ώρα σας και θα σας παρακαλούσα να αρχίσετε με το παρουσιάζοντας το ε, Ευρωπαϊκό Πιλωτικό Πρόγραμμα για το Alzheimer και να ξεκινήσουμε μετά τη συζήτηση. Η κυρία Ντράγκια Άκλη έχετε το λόγο. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την, την παρουσίαση, την εισαγωγή που κάνατε και χαίρομαι που είσαστε εδώ τόσο νωρίς για να ακούσετε για το κοινό μας πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και ιδίως για το Alzheimer. Θα ε, ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι στις 22 Ιουλίου φέτος ε, η Κομισιόν υιοθέτησε μια πρόταση για μια σύσταση του Συμβουλίου για μέτρα καταπολέμησης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, ιδίως του Αλτσάιμερ μέσω ενός κοινού προγράμματος. Η σύσταση αυτή καλεί τα κράτη-μέλη να εδραιώσουν καταρχάς ένα κοινό όραμα για το πώς θα αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταλάβουμε, εντοπίσουμε, προλαμβάνουμε και καταπολεμήσουμε νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Επίσης, για να καθιερώσουμε, για να φτιάξουμε ή δημιουργήσουμε μία στρατηγική ερευνητική ατζέντα ε, η οποία θα ορίζει τις έρευνες, τις αναγκαίες έρευνες που πρέπει να γίνουν και τρίτον να ε, ε, αναπτύξουμε μία, ένα πλαίσιο διαχείρισης του όλου θέματος. Γιατί λοιπόν επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και δει το Alzheimer. Καταρχάς, πρέπει να πούμε γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ασθένεια. Είναι ένα από τα θέματα προτεραιότητας στην, ε, της υγείας, στον του, τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πάρα πολύ ε, γρήγορα αναπτυσσόμενη ασθένεια και βλέπετε του πίνακα εδώ πώς εξελίσσεται η ασθένεια της άνοιας, ε, της του Πάρκινσον και του, ε, της εμβολής. Είναι λοιπόν το Alzheimer ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας στην Ευρώπη και ένα μεγάλο πρόβλημα διεθνώς. Βλέπετε ακριβώς εδώ στον πίνακα τα στοιχεία, τον αριθμό των ανθρώπων ε, που θα προσβληθούν από εκφυλιστικές ασθένειες, άνοια και Alzheimer. Σήμερα 35,6 εκατομμύριο, ενώ σε 40 χρόνια 115,4 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν τη ραγδαία άνοδο των ανθρώπων που θα έχουν προσβληθεί. Η, το Alzheimer είναι η πιο κοινή νευροεκφυλιστική ασθένεια <clears throat> και αντιπροσωπεύει το 50-70% όλων των εκφυλιστικών των ανιών στην Ευρώπη είναι ο τέταρτος πιο κοινός παράγοντας παγκοσμίω εκφυλιστικών ασθενειών. Εμένοντας τους αριθμούς, βλέπετε εδώ ότι 7,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν από Alzheimer και διάφορες ε, συγγενείς ε, μορφές ε, άνοιας, δηλαδή 12,5 Ευρωπαίοι ανά χίλιους αυτές δεν είναι ε, ε, After the initial diagnosis. Δεν είναι ασθένειες που οδηγούν αναγκαστικά στο θάνατο, αλλά οι άνθρωποι μπορεί ε, να ζήσουν, αλλά να χειροτερεύουν σταδιακά για 7 με 12 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση. Υπολογίζουμε ότι περίπου 19 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θίγονται ε, καθημερινά από αυτήν την ασθένεια, δεδομένου ότι ε, έχει άμεση επίπτωση στους γενικό και κονιακό περιβάλλον. Τελικά οι περιπτώσεις οι οποίες, ε, ο ρυθμός ο οποίος εμπλέκεται στο όλο πλαίσιο των, περιπτώσεων και επιπτώσεων του Alzheimer είναι περίπου 100, είναι το 2005, το κόστος δηλαδή ήταν 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί λοιπόν πρέπει να, προσέ... να δώσουμε τόση προσοχή στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και ιδίως το Alzheimer. Είναι ένα τομέα προτεραιότητα, όπω σα είπα, επειδή είναι τόσο ε, ε, εξέχουσα περίπτωση <clears throat> στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ολοκληρωμένη ε, τακτική, προστατηγική έρευνα και να τη χρηματοδοτήσουμε. Είναι μια προτεραιότητα αυτή την οποία πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε. Το 2005 οι συνολικές δαπάνες για έρευνες των εγκέφαλων στην Ευρώπη ήταν 4,1 δις ευρώ και από αυτά 855 εκατομμύρια προήλθαν από τον δημόσιο κορβανά. Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πλαίσιο και τα προγράμματά του δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο Alzheimer και έχουν διαθέσει 136 εκατομμύρια ευρώ από το 2002 μέχρι το 2006 και 102 εκατομμύρια έχουν <clears throat> δοθεί, ε, ε, ε, έχουν δαπανηθεί για αυτό τον σκοπό, θα δοθούν μάλλον το 2007-2009. Το 1 τρίτο δηλαδή όλων των επενδύσεων, όλων των κονδυλίων που διατίθεται για έρευνε του εγκεφάλου. Είναι λοιπόν, όπως σας είπα, ένα, ένα πρόβλημα προτεραιότητος, το οποίο χρειάζεται εμπεριστατωμένη και ε, εκτεταμένη έρευνα. Δεν ξέρουμε γιατί χρειάζεται αυτή η έρευνα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα ε, από, γιατί ε, εκδηλώνεται το άτσαμα και δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία είτε να, για να σταματήσει είτε να βελτιώσει την κατάσταση των ασθενών. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυτάρων. Είναι επίσης και παράγοντες κινδύνου δεν έχουν εντοπιστεί. Η διάγνωση και επίσης πάρα πολλές περιπτώσεις δεν διαγνώσκονται. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μία ουσιαστική έρευνα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε, να καθορίσουμε και να μελετήσουμε όλους τους παράγοντες που που οδηγούν ε, στο Alzheimer για να εφαρμόσουμε μια προληπτική τακτική, να κάνουμε μια σωστή διάγνωση και να μπορέσουμε να προλάβουμε την εκδήλωση της, της ασθένειας. Ε, δεν έχει νόημα <clears throat> να καταλήξουμε σε ερευνητικά αποτελέσματα 50 χρόνια μετά την εκδήλωση της, ε, των συμπτωμάτων. Πρέπει όλα αυτά να τα ε, εντοπίσουμε και να τα ορίσουμε ε, πολύ νωρίτερα, προληπτικά δηλαδή. Σε ποιους τομείς τώρα χρειάζεται να γίνει έρευνα. Εάν συγκρίνεται το Alzheimer που είναι η μικρή κόκκινη ε, κουκίδα στο κάτω αριστερά παρελόγραμμο, έχετε μία πολύ χαμηλό δίκτυ ερευνητικού συντονισμού ενώ επάνω δεξιά υπάρχει υψηλός ερευνητικός ε, συντονισμός για άλλες ασθένειες και ε, γι' αυτό επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η διάσπαση ε, της έρευνας πρέπει να τη συντονίσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε έναν καλύτερο συντονισμό και να συγκεράσουμε όλες τις προσπάθειες. Ποια θα είναι λοιπόν τα αποτελέσματα η ευρωπαϊκή εικόνα είναι διασπασμένη και διάχυτη διότι υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης ερευνητικών πολιτικών και οργανωτικών δομών στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία αδύναμη διασύνδεση μεταξύ των βασικών ε, κλινικών και δημοσίων ερευνητικών προγραμμάτων και έτσι δεν μπορούμε να συγκεράσουμε όλη αυτή τη γνώση και την εφαρμόσουμε πρακτικά έτσι ώστε να ωφεληθεί η θεραπεία και η φροντίδα. Χρειάζεται λοιπόν ένα συντονισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος θα επιτρέψει μια κρίσιμη μάζα δεξιοτήτων, γνώσεων και πόρων να συγκεραστούν για να μπορέσουν να συντονίσουν ε, και να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις της ε, ασθένειας. Πώς θα εφαρμόσουμε λοιπόν αυτή την πιλωτική πρωτοβουλία κατά πολέμησης νευροεκφυλιστικών ασθενειών και δι του Alzheimer αν ε, το δείτε όλη αυτή την προσπάθεια μέσα σε ένα πλαίσιο, θα οργανώσουμε έναν κοινό προγραμματισμό βάσει της ανακοίνωσης της Κομισιόν που έγινε τον Ιούλιο του 2008 και της απόφασης Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 η οποία ε, λέει ότι τα κράτη-μέλη προαιρετικά και επί τη βάση μιας ε, κειμενόμενης γεωμετρίας ε, θα ασχοληθούν με τον ορισμό ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής ατζέντα για την έρευνα η οποία θα βασίζεται στο κοινό όραμα και θα αντιμετωπίζει τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Αυτό το κοινό πρόγραμμα λοιπόν θα μεγιστοποιήσει την αξία των εθνικών επενδύσεων στην έρευνα για το, το Alzheimer, θα ενισχύσει το συντονισμό των εθνικών ερευνητικών προσπαθειών σε αυτό τον τομέα, θα μειώσει τους φραγμούς και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στον, ε, στον συντονισμό της έρευνας και, στην, ε, και στη διάσπαση των ερευνητικών ε, προσπαθειών θα ενισχύσει τους βασικούς δεσμούς ε, και σχέσεις μεταξύ της βασικής κλινικής και κοινωνικής έρευνας και θα επιταχύνει τη διάχυση της βασικής γνώσης σε αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Brain. Αν δείτε λοιπόν το yes, τον υγιή, έναν υγιή εγκέφαλο και έναν εγκέφαλο που έχει προσβληθεί από τον Alzheimer και έχει συρρυκνωθεί και εκφυλιστεί, βλέπετε τη διαφορά. Ε, προφανώς λοιπόν χρειάζεται να γίνει αυτό το κοινό πρόγραμμα για να ε, αναπτύξουμε νέες μας θεραπευτικές μεθόδους, να αξιολογήσουμε τους ε, παράγοντες κινδύνου, να μελετήσουμε την, τον, τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν σε πληθυσμιακές ομάδες, να τυποποιήσουμε τα διαγνωστικά κριτήρια και τα ε, ε, ε, μέσα αξιολόγησης. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία του κοινού προγράμματος. Το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2008 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών αναγνώρισε τις προκλήσεις που παρουσιάζουν από αυτή την ανάπτυξη των ευρωεκφυλιστικών ασθενειών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να ε, συντονιστεί ε, να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε όλα τα κράτη-μέλη όπου, η οποία θα υποστηριχθεί από την Κομισιόν και τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο τη μείωση της εμφάνισης των ασθενειών αυτών. Και υιοθετήθηκε αυτή η πρόταση ε, του Συμβουλίου το 25 Σεπτεμβρίου 2009 στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Αυτή τη στιγμή 20 κράτη-μέλη συζητούν τις διάφορες μορφές και πτυχές ε, αυτού του προγράμματος ε, που χρειάζονται για την ε, εδραίωση αυτής της πρωτοβουλίας. Η Κομισιόν θα συμβάλλει προσφέροντας από το 2010 ένα πλαίσιο χρηματοδοτικό και νομικό για την υποστήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη της στρατηγικής ερευνητικής ατζέντα και η πρωτοβουλία αυτή ε, θα συμπληρώσει άλλες προσπάθειες που γίνεται μέσα στην ε, κοινότητα, παράπλευρες προσπάθειες και θα έχει τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Alzheimer και άλλες ε, εκφυλιστικές ασθένειες, άνοιες». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει πολλές φορές ε, δείξει και εκδηλώσει το ενδιαφέρον του ε, και επίσης ότι την κατανόησή του για τη σημασία που έχει η έρευνα του Alzheimer για τους Ευρωπαίους πολίτες και υποστηρίζει πλήρως αυτή την προσπάθεια και στη γνωμοδότησή του κοινό πρόγραμμα πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή χαιρετίζει αυτή την προσπάθεια, αυτή την πρωτοβουλία. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ εκτενής ε, και πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Και τώρα καλό θα ήταν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Ο κύριος Λάμπερς που είναι εισηγητής έχει πρώτος το λόγο. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεν το συνηθίζω και θα προσπαθήσω στο μέλλον να το αποφεύγω. Δεύτερον, είναι η πρώτη μου έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξή. Το πιθανότερο χρειαστώ τη βοήθειά σα και από τη Γραμματεία και ε, των συναδέλφων για να ε, βεβαιωθούμε ότι θα είναι χρήσιμη η έκθεση. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα μερικέ σκέψει ε, καθώ μπαίνω στην έκθεσή μου. Για το θέμα αυτό το Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει. Δεν είναι στη συναπόφαση το θέμα. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε όλη τη διαδικασία. Να υπάρξει μια προστιθέμενη αξία. Αντί να καθόμαστε στην άκρη και να επικρίνουμε απ' έξω αυτά που συμβαίνουν. Για μένα αυτό τι σημαίνει λοιπόν, που μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο. Πρώτον, για το τι πρόκειται να κάνουμε. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε όταν μιλάμε για νευροεκφυλιστικά νοσήματα δεν ασχολούμαστε μόνο με την όσο Αλσχάιμερ, το σύνολο των νοσημάτων. Και επίσης να βεβαιωθούμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο ε, η θεραπεία της νόσου, αλλά και η αντιμετώπιση των αιτιολογικών ε, καταστάσεων. Δηλαδή εντάξει, να κάνουμε ε, καλά τους ασθενείς, αλλά να μειώσουμε ε, ιστοδύνικες τον αριθμό των ε, ανθρώπων που αρρωσταίνουν. Να καταλάβουμε δηλαδή την αιτιολογία της νόσου για να την πολεμήσουμε στη ρίζα της. Αυτά είναι τα δύο σκέλη της εξίσωσης. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι το, το, το πώς. Είπαμε το τι, τώρα πάμε στο πώς. Δεν ξέρω τι γίνεται με το κοινό πρόγραμμα. Κατάλαβα ότι είναι μια πρωτοβουλία. Εγώ είμαι καινούριο στα θεσμικά όργανα. Έχουμε την εντύπωση απ' έξω ότι είναι πολύ καλή ένωση στο να δημιουργεί νέα εργαλεία, νέους οργανισμούς, ε, νέους θεσμούς, νέες μεθόδους. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ρεαλιστές στην προσέγγιση μας και πρακτικοί θα κάνουμε το πρόγραμμα αυτό, είπαμε το κοινό, αλλά πώς θα πρέπει να συγκλίνουν οι προσπάθειές μας και να έχουμε και αποτέλεσμα. Δηλαδή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε αντί να προσθέτουμε νέους θεσμούς και όργανα. Δεν ξέρω αν στον αστερισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση υπάρχουν θεσμικά όργανα ή άλλα όργανα ήδη υπάρχοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω φορέα αυτή τη συνεργασία πάντω ε, θα ρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει πολύ και απλώ όχι να ερχόμαστε να προσθέτουμε και νέε δομέ. Κάποιε πρώτε σκέψει ήταν αυτέ σε πρώιμο στάδιο και βλέπω εδώ του και ηγητέ που είναι παρόντε, Μίλησα και με άλλου εχθέ. Θα προσπαθήσω να επιβεβαιώσω σύντομα να συγκαλέσω μια πρώτη συνεδρίαση των σχεδόν ε, εισηγητών για να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σουρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω ε, ότι θα έχει πολύ ισχυρά ε, έτσι και κοινωνική επίπτωση γιατί δεν ε, υποφέρουν μόνο οι ασθενείς αλλά και ο περίγυρος ο οικογενειακός και εμείς πηγαίνουμε συχνά σε οίκους ευγυρίας και βλέπουμε πως έχει νόσο στο τελικό στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε λίγο περισσότερο γιατί προκύπτει, πώς ε, προκύπτει αυτή η ασθένεια, πώς μπορούμε να την ε, αποφύγουμε ή να τη θεραπεύσουμε. Υπάρχει στο εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι μια επιτροπή επιστημονική που ασχολείται με αυτά τα θέματα, με την επιστημονική πλαισίωση της τεχνικής νομοθεσίας και είχαμε πολλούς ε, επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη του εγκεφάλου και μάθαμε ότι μπορεί να μεταξελιχθεί ο εγκέφαλος. Λοιπόν, ερώτηση υπάρχουν τομείς σε αυτό το κλάδο της επιστήμης και της έρευνας ε, που να ασχολείται κάποιος με αυτό πώς ε, προάγεται η λειτουργία και η ανάπτυξη του εγκεφάλου και σε προχωρημένη ηλικία πώς μπορεί να ερεθιστεί αυτή η διαδικασία για να έχουμε αναπαραγωγή, ανανέωση του εγκεφάλου. Έχουν γίνει ήδη πολλές ε, συζητήσεις εδώ για τη βιοτεχνολογία, για τα βλαστικά κύτταρα. Τι θα γίνει λοιπόν Τι γίνεται με την έρευνα ε, του εγκεφάλου και έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 136 εκατομμύρια. Πού είναι η καρπή αυτών των ερευνών και στην ανάλυση του 7ου προγράμματος πλαισίου συμπεριλαμβάνεται αυτό και πώς φαντάζεστε εσείς στη συνέχεια στο 8ο πλέον ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανίστερ Ρόι. φανιστερ Πρόεδρε. από την παρουσίαση που ακούσαμε και σήμερα από την νέα διευθύντρια, σημείωσα ιδιαίτερα και κοίταξε ιδιαίτερα το γράφημα αυτό που λέτε ποια είναι η ένταση της έρευνας στην Ευρώπη και τι κάνουμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι. Και βλέπουμε όλες αυτές τις κουκίδες και τελικά ε, υπολείπεται η έρευνα του εγκεφάλου. Λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα ε, και μας ενδιαφέρει πολύ, αλλά έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το σημαντικό τομέα. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των κρατών μελών κτλ. Έχω όμως την εξή ερώτηση. Από τη μια έχετε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με σαφή κατεύθυνση και τώρα λέτε ένα νέο ε, εργαλείο αυτού του κοινού προγραμματισμού. Και τι θα γίνει, α πούμε, σε δύο-τρία χρόνια τι θα κάνουμε. Η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ε, δαπανίσει περισσότερο, να επενδύσει περισσότερο και από το πρόγραμμα πλαίσιο και να δώσει κάποια καθοδήγηση. Ε, και στην έρευνα. Καλές είναι οι καλές πρωτοβουλίες, αλλά τι να το κάνω να είμαστε με 20 ε, ε, άλλους εταίρους σε ένα καράβι και να προσπαθούμε να πάμε κάπου όλοι μαζί, χωρίς να ξέρουμε πού είναι αυτό. Και ποια είναι η ιδέα σα εσείς τι προτείνετε με βάση αυτό το γράφημα που μας δείξατε. Και σε σχέση με τα όσα είπε και ο εισηγητή, με ενδιαφέρει να δούμε τι ρόλο παίζει το Κοινοβούλιο. Εγώ δηλαδή είμαι εδώ πέντε χρόνια, ποτέ δεν το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε ότι 90% ε, του προϋπολογισμού για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι από τα κράτη-μέλη. Ε, εκτελείται δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Και ε, ποιε είναι οι δεσμεύσει, ποιο είναι ο προπολογισμό που έχουμε τώρα. Ακούσαμε ότι υπάρχουν 136 εκατομμύρια, αλλά σε σχέση με τα καρδιαγιακά νοσήματα και τον καρκίνο είναι μικρό το ποσό και σημαντικά μικρότερο. Και σιγά σιγά, επειδή αρχίζουμε να αναλύουμε και να αξιολογούμε το 7ο πρόγραμμα για να περάσουμε στο επόμενο, θα πρέπει να μας απασχολούν αυτά τα θέματα. Ε, η δική μας σκιώδη συγκήτρια λείπει, είναι η κυρία Κροστέτ. Ε, το έφεραν οι Γάλλοι αυτό που βιαζόντουσαν κιόλα πολύ στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό θέμα στην κοινωνία και απασχολεί και τον κόσμο και το δικό μας. Ε, και θα καλό να δώσουμε μια κατεύθυνση και στην έρευνα. Ευχαριστώ πολύ και να μας πείτε πώς να κάνουμε τις τροπολογίες μας για να βοηθήσουμε και εμείς αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή συμπληρώση και συμπληρωματική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Θα με ενδιαφέρει και εμένα να μου πείτε λίγο τα μεγέθη, τα οικονομικά, έτσι, και σε σχέση με άλλες ασθένειε ακριβώς. Η κυρία Γκουτιέρης Κορτίνες. Muchas gracias, señor Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπαν προσαντλήσαντες και δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο από όλα αυτά που ακούσαμε και θέλω να ρωτήσω την κυρία Γενική Διευθύντρια. Για ποιους λόγους πιστεύετε εσείς ότι στην Ευρώπη, πώς να το πω, είναι χαμηλή αυτή η δυνατότητα να κάνουμε το θέμα αυτό προτεραιότητα. Τι έγινε, δεν έχουμε ερευνητέ. Έχουν έρθει ενώσει και σωματεία και ενώσει επιστημόνων εννοώ και ερευνητών που ε, παραπονιούνται και διαμαρτύρονται ότι δεν του αναγνωρίζουν. Ή υπάρχουν άλλοι λόγοι γιατί συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Και ένα δεύτερο. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το Κοινοβούλιο να δοθούν κίνητρα και ε, οικονομικά είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Γιατί πραγματικά ε, μας εκλυπαρούν αυτές οι οικογένειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας και συγχαρητήρια που έχετε θέσει αυτό το κέντρο βάρους. Ο Πάουλ Ρούμπιχ είπε προηγουμένως ότι το Κοινοβούλιο έχει την Επιτροπή ΣΤΟΑ ε, και ακριβώς ε, ε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για τις ασθένειες του εγκεφάλου. Όλα αυτά τα καλωσορίζουμε. Αλλά, και έρχομαι στο αλλά τώρα, ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Μα η πόρη εδώ είναι από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο και έπεται σύντομα το 8ο. Μου κάνει εντύπωση ότι στο παράδειγμα της νόσου Alzheimer που είναι μια ασθένεια που αφορά όλη την κοινωνία και τη διαπερνά οριζόντια. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν ακόμα ε, αλληλοεπικαλύψεις, δίπλες έρευνες και υπερβολική γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει αυτό. Ακούστηκαν τα 136 εκατομμύρια ευρώ. Ε, καλά δεν είναι και τίποτα τρελά λεφτά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι περιορισμένο το ποσό, αλλά ε, όσο και να είναι, είναι χρήματα των φορολογουμένων και έχουμε διπλή έρευνα και κακό συντονισμό. Αυτό έχει να κάνει με ματαιοδοξίες κρατών, με ματαιοδοξίες έρευνητών και νομίζω ότι αυτό το νόσημα ακριβώ δείχνει ότι μας αφορά όλους, ότι αναπτύσσεται και αυξάνεται και πολύ ωραία τα είπατε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε επιγόντω να καταπολεμηθεί, γιατί δεν ξέρουμε σε τι οφείλεται. Λοιπόν, θα ήταν εδώ ένα καλό παράδειγμα για να οξύνουμε, να κατευθύνουμε περισσότερο την έρευνα προς τα εκεί και να αφαιρέσουμε τη γραφειοκρατία. Αυτή είναι η μεγάλη δουλειά του Κοινοβουλίου στο 8ο πλέον πρόγραμμα πλαίσιο και σε σχέση με αυτά που είπε η συνάδελφος μόλις, δικό μας όπλο και εργαλείο είναι ο προπολογισμό. Βεβαίως θα συνεργαστούμε αλλά θα τρίξουμε λίγο και τα δόντια αν χρειάζεται να περιορίσουμε τα κονδύλια για να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Κατά τα άλλα υπάρχουν και ιδιωτικέ, ξέρετε, πρωτοβουλίες που ασχολούνται με την νόσο Alzheimer. Ξέρω ότι το 7ο πρόγραμμα, όπως και το 6ο, είναι ανοιχτό για την ιδιωτική συμμετοχή, αλλά ξέρουμε ότι θα πρέπει να φτιάξουν ομίλου. κάποιο που δεν είναι μέσα και παρόλα αυτά ασχολείται με την ε, Alzheimer δεν φτάνει στα κονδύλια. Λοιπόν, θα πρέπει να τα ανοίξουμε και ε, περισσότερο για ιδιωτική πρωτοβουλία. Κυρίες και κύριοι, εδώ χρειάζεται τώρα ε, ριζική αλλαγή. Να πάρουμε αυτή την όσο και να πούμε εμείς. Οι Ευρωπαίοι θέλουμε να ε, προχωρήσουμε τώρα σε καμπή. Και το πρώτο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η πρόληψη. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να προληφθεί η νόσος. Δεν τα ξέρουμε, υπάρχουν κάποιες συγκεχημένε πρώτε ιδέες. Αυτό θα πρέπει να είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν ακόμα προσβληθεί από την νόσο να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Στο διαβήτη το ξέρουμε, το καταφέραμε με κίνηση, σωματική άσκηση, με διατροφή, γιατί είναι μεγάλο νόσημα μαζικό. Μέτρα ε, λοιπόν προληπτικά στον καρκίνο του παχαίου σαντέρου επίσης το γνωρίζουμε πολύ νωρίς, υπάρχει η πρόνοια και η πρόληψη, αλλά στην Αλσχάιμερ αυτό το αγνοούμε. Και να πω και κάτι άλλο τώρα για τα αποτελέσματα. Το ζούμε στη ΣΤΟΑ με το Ρούμπιχ και με άλλους συναδέλφους. Τα αποτελέσματα συχνά ε, είναι ε, προστατευμένα από ε, διπλώματα ευρυσιτεχνίας. Και εμείς οι Ευρωπαίοι μετά έρχομαστε σε μια δινή θέση και παρακαλώ την Κομισιό να το σκεφτεί. Μήπως θα πρέπει ως υπόδειγμα να χρησιμοποιηθεί η νόσος Alzheimer για να κοιτάξουμε τα θέματα των ευρεσιτεχνιών στη δημόσια υγεία. Να το ξανασκεφτούμε. Μπορεί να χρειάζονται μόνο γιατί αυτό είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό εμποδίζει ε, και ε, ε, δεν βοηθάει την έρευνα. Alzheimer και στο λεγόμενο evergreening έχουμε αυτά τα προβλήματα. Να το σκεφτούμε, να ε, το κοιτάξουμε για να προχωρήσουμε και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και τελευταίο. Οι βιολογικές επιστήμες προσφέρονται εκτός από την έρευνα για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής για να ξανάρθουμε ε, στην αιχμή της έρευνας οι Ευρωπαίοι και προσφέρεται ακριβώς η Alzheimer για να ενώσουμε επιτέλους τις δραστηριότητες μας οι Ευρωπαίοι και να δείξουμε ότι δεν είμαστε τόσο κακοί όσο μας θέλει η φήμη μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντιπρόεδρος, η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ την ε, δόκτωρα Ντράγκια για την παρουσίαση που μας έκανε. Μελέτησα το έγγραφο αυτό όπως και την προηγούμενη ανακοίνωση της Κομισιόν, με ορισμένους επιστήμονες στην Ιταλία και δηλώνω ότι η σύσταση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα. Σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση, όπως την έκριναν τα άτομα αυτά που δουλεύουν σε κέντρα αριστείας επιστήμονες, δηλαδή το περιεχόμενο αυτής εδώ της ανακοίνωσης που είναι η μετάφραση κατά κάποιο κοινού προγραμματισμού κρίνεται θετική και δείχνει μια ψηλό επίπεδο επιστημονικής συνειδητοποίησης των μεγάλων θεμάτων έρευνας που σχετίζονται με τα νευροεκφυγιστικά νοσήματα και συγκεκριμένα το Αλσχάμερ. Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής δύο τεινά. Με βάση αυτά που ακούσαμε και που επανάλαβαν και πολλοί συνάδελφοι, φαίνεται ότι στον τομέα αυτό το σημαντικό είναι να ξεπεραστεί ο σημερινός κατακαιρματισμός. Η δυσκολία της έρευνας για να εντοπίσει τα αίτια αυτής της νόσου, του εκφυλισμού δηλαδή των ε, εγκεφαλικών κυτάρων, απαιτεί συγκέντρωση. Λίγα μεγάλα προγράμματα όπως γίνεται στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη ΣΥΠΑ, δηλαδή εκεί όπου κυβερνήσει και ιδιωτικέ εταιρείε χρηματοδοτούν τεράστια προγράμματα με πάρα πολλού πόρου για συγκέντρωση στην έρευνα με δείκτε και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί μια φαρμακευτική θεραπεία. Η Ευρώπη λοιπόν, πέρα από το ότι να τονίσει αυτή την ανάγκη συντονισμού της έρευνας μας και των κρατών μας. Πώς μπορεί να ευνοήσει, να βοηθήσει αυτό το συντονισμό, αυτή τη συγκέντρωση που σημαίνει να μπουν οι πόροι από κοινού σε κοινά ορισμένα, από κοινού ορισμένα προγράμματα. Και το δεύτερο ερώτημα. Προβλέπετε κάποια μορφή επιστημονικής συνεργασίας και συντονισμού μέχρι ότου να φτάσουμε σε διπλώματα τεχνίας. Και έχω κατά νου αυτό που γίνεται στην Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ιαπωνία όσον αφορά την νόσο αυτή. Ειδικά για την Ευρώπη. Πώς μπορούμε να πείσουμε τις κυβερνήσεις τα λίγα κέντρα αριστείας που λειτουργούν σε σχέση με το πρόβλημα αυτό να συνεργαστούν και για έρευνα και για θεραπεία. Πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα. Θα έπρεπε εντό εισαγωγικών να, υποχ... να τους υποχρεώσουμε να συνεργαστούν. Διαφορετικά οι λιγοστοί πόροι δεν θα αποδώσουν. Και μία τελευταία παρατήρηση. προκειμένου να υπάρχει ένα όργανο για την αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εγώ όταν ακούω για νέα όργανα πάντα ανησυχώ γιατί θεωρώ ότι μάλλον θα βαρύνουν στο σύστημα γραφειοκρατικά και ως, όσον αφορά το κόστος. Να μην δημιουργήσουμε μια νέα υπηρεσία, ένα νέο θεσμό, ένα νέο όργανο που υπάρχει κίνδυνος αντί να βοηθήσει να αποτελέσει βάρος. Επαναλαμβάνω όμως, ε, θεωρώ θετικά τα μέχρι τώρα προτινόμενα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα, διότι πολλά από εκείνα που θα ήθελα να πω τα είπαν οι συνάδελφοί μου και με κάλυψαν. Καταρχά, θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω για τι εξηγήσει σα, πολύ ενδιαφέρουσε και πολύ σαφεί, κυρία Γενική Διευθύντρια. Αυτά που μας είπατε μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ για τα εξή δύο. Ε, πρώτο από το θέμα το ίδιο, το είπαν ξεκάθαρα οι συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα από επιστημονικής πλευράς και δεν θα μπω ε, σε λεπτομέρειες γιατί πλέον δεν είμαι και ειδική σε αυτά τα θέματα αλλά μπορώ να σας πω ότι σήμερα γνωρίζω λίγο περισσότερα μετά από αυτά που μας είπατε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να γνωρίζουμε λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να παίρνουμε πολλές πολιτικές αποφάσεις και σε ένα τέτοιο θέμα πολύ περισσότερο. Και είναι και πάρα πολύ επίμαχο το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. αν Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έρευνα, ε, όθηση και ενίσχυση στην έρευνα σε βλαστοκύτταρα ή όχι. Ε, και σας ευχαριστώ. Έρχομαι στο δεύτερο ε, αίτιο, γιατί μας ενδιαφέρει λοιπόν. Διότι ακριβώς ε, ε, φτιάξατε ένα νέο μέσο ενίσχυσης της έρευνας και θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, καταλαβαίνω ότι φιλοδοξείτε να απαντήσετε σε ένα από τα προβλήματα που ανέκαθεν ναι, θέτουμε εμείς που είναι ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών προγραμμάτων και μεταξύ των κρατών μελών ο συντονισμός χωλαίνει. Από ό,τι φαίνεται είναι το καλό μέσο αυτό εργαλείο. Επίσης έχω καταλάβει ότι επιλέξατε αυτό το θέμα ως πιλωτικό πρόγραμμα διότι είναι ένα θέμα πραγματικά ε, στο οποίο έχονται και πολλά κρατημέλη αλλά και δίνουν πολλά χρήματα σε αυτή την έρευνα. Λοιπόν, προσφέρετε το θέμα δηλαδή για να ε, προσπαθήσει κανείς να φτάσει στο συντονισμό. Έρχομαι τώρα στις συγκεκριμένες με ερωτήσεις που θα ήθελα παρακαλώ να με διαφωτίσετε λίγο παραπάνω. Γιατί επιλέξατε τελικά αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο, τι φέρνει, τι προσφέρει που δεν επρόσφεραν τα προηγούμενα βάσει του άρθρου 169. Επίσης θα ήξερα να γνωρίσω λίγο περισσότερο για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσείς ε, λανσάρατε και προωθείτε αυτή την ε, προσπάθεια συντονισμού, αλλά ο δικός σας ρόλος ποιος θα είναι. Και αυτό είναι σημαντικό για να ορίσουμε και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να μπω σε αυτό, το είπαν οι συνάδελφοί μου. Καταρχάς, ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Και δεν μας αρέσει αυτό στην Επιτροπή μας. Αλλά θα θέλαμε λίγο περισσότερο να μας πείτε ε, τις προθέσεις σας, τους στόχους σας και μπορεί να έχετε πολύ το δίκιο. Ένα άλλο ερώτημα. Προσπαθήσατε, βολιδοσκοπήσατε τα κράτη-μέλη, ξέρετε πώς αντιδρούν, ε, πώς απαντούν, δέχονται αυτό το νέο μέσο, τι, τι, πώς το βλέπουν, πώς το αξιολογούν. Και επίσης, έχετε προγραμματίσει το, τι θα γίνει με τα αποτελέσματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, πώς θα γίνει η ε, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επίσης μας είπατε σαφώς ότι πρόκειται για ένα, ένα θέμα διεπιστημονικό. Και σας ερωτώ, γιατί δεν προκηρύξατε κοινό ε, διαγωνισμό όπως προβλέπετε σε ένα τέτοιο πλαίσιο με νέες τεχνολογίες για τη διάγνωση, προφανώς έρευνα, ε, θέματα υγείας κτλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο, ο συνάδελφος Τζιπ έχει το λόγο, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σωστό, σωστά είπατε το όνομά μου. Θα ήθελα να... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα είναι αυτό που είπατε για το συντονισμό κοινωνικής έρευνας και κλινικών πειραμάτων. αυτή η πρωτοβουλία που θα βοηθήσει και τις οικογένειες και αυτές που περιθάλπουν γενικά άτομα που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους θα έχει επίπτωση στη ζωή 19 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ένα παράδειγμα της θετικής επίπτωσης που μπορεί να έχουν κοινέ πολιτικές. Στο Ευρωκοινοβούλιο όλοι μας νομίζω πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη συντονισμού και της έρευνας και των προσπαθειών και των πόρων. Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ένωσης για να συντονιστούν όλα αυτά. Οι Ευρωπαίοι σίγουρα είναι υπέρα μια τέτοιας κίνησης. Στη χώρα μου, την Πολωνία, η νόσος αυτή αυξάνει συνεχώς. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, άρα υπόκεινται όλο και περισσότερο στον κίνδυνο αυτής της νόσου. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα για τις οικογένειες και βλέπουμε ενώσεις οικογενειών και ατόμων που περιθάλπουν τους νοσούντες να αυξάνονται σε όλη τη χώρα. Αυτό όμως δεν λύνει το βασικό πρόβλημα. Πώς να προλάβουμε και να θεραπεύσουμε την νόσο αυτή. Πώς να γίνει έρευνα έτσι ώστε να βελτιωθεί η θεραπεία. Από ό,τι έχω καταλάβει από αυτό που μας είπατε στην ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Όλες οι χώρες της Ένωσης ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα αυτό. Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν αυτό το κατάλαβα σωστά. Και έχω και ένα ερώτημα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα κοινωνικά και κλινικά πειράματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εξίσου από την Ένωση ή τα κλινικά πειράματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται περισσότερο από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και όχι από την Ένωση. Ευχαριστώ τελευταίο ο κύριο Σόσα Βάγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα, διότι τώρα πια η συζήτηση ξεκαθαρίζει. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω το εξής και μόνο το απλό γεγονός ότι συζητάμε για το θέμα αυτό εδώ ε, δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, διότι η Ευρώπη, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να δείχνουν πολύ μεγάλη ευαισθησία και το γεγονό, λοιπόν και μόνο ότι το συζητούμε εδώ θα πρέπει να είναι για όλους μεγάλη ικανοποίηση. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, ο ρόλος της Ευρώπης, ο ρόλος των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι η προώθηση και ενίσχυση της έρευνας στο θέμα αυτό. Αυτό και μόνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και θέση σε μια αρχή που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, που είναι η αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών ή περιφερειών στην Ευρώπη, για να μην πω και σε δήμους και κοινότητες, να γίνεται επιτόπου. Οπότε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων θα πρέπει αποκλειστικά να στρέφεται στο να υποστηρίζει την υψηλή έρευνα την υψηλή έρευνα στα κράτη-μέλη. Και ένα τελευταίο κάτι που υπόθηκε κάποια στιγμή εδώ, που είναι η ανάγκη να μην δημιουργούμε, ή να το πω να αποφεύγουμε όσο γίνεται τη δημιουργία νέων διοικητικών και γραφειοκρατικών δομών. Αυτό είναι ένα θέμα που επανέρχεται συχνά. Μία από τις ε, επικρίσεις που ακούμε και τις αιτιάσεις και τις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων πολιτών είναι ότι έχουμε πολύ πυκνό ε, ε, οργανόγραμμα και πάρα πολύ βαρύ, έτσι, μπαρόκ ε, να ενισχύσουμε την έρευνα λοιπόν και να αναδείξουμε και πάλι την αρχή της ε, επικουρικότητας που είναι βασική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και θα δώσω το λόγο ε, στην ε, κυρία Διευθύντρια να απαντήσει στις ερωτήσεις και στα σχόλια ε, σύντομα. ελπίζω να τα καταφέρετε. Μπορώ και μιλώ ταχύτατα. Έχω... Θα απαντήσω σε τρία μέρη. Καταρχάς τις ερωτήσεις που αφορούν την έρευνα και πράγματι Χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε όλα τα επίπεδα, αρχίζοντας από τη βασική έρευνα που καλύπτει ε, τις ε, μεθόδους από την ε, κανονική διαδικασία ε, έως τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες για να μπορούμε να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό των, ε, της κλινικής και της βασικής, μεταξύ κλινικής και βασικής έρευνας. Άρα δεν χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθεί μόνο ένας τομέας, διότι είναι αλληλένδετη αυτή η ερευνητική τιμή, άρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ε, ουσιαστική στρατηγική από την ε, πρόληψη στη διάγνωση και στη θεραπεία υπάρχουν, υπάρχει σαφώς ανάγκη συντονισμού της ε, καλής έρευνας, της ε, υψηλής έρευνας, διότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται τεχνικές ε, και μέθοδοι οι οποίες είναι πολύ δαπανηρές και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι στις προσπάθειες συντονισμού που έχουμε κάνει Προσπαθούμε ακριβώς να εντοπίσουμε ε, ποιες είναι οι έρευνες που μας ενδιαφέρουν, πού γίνονται και σε τι κλάδους, ε, σε, σε ποιο συγκεκριμένο αντικείμενο γίνονται αυτές οι έρευνες. Άρα λοιπόν σαφώς χρειάζεται συντονισμός και εντοπισμός του τι περισσότερο χρειάζεται να γίνει. Εάν τώρα μελετήσουμε το όφελος και πώς το όφελος αυτό θα αγγίξει τον ασθενή είναι σαφές ότι και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι πολλές ε, ε, φαρμακευτικές εταιρείες μέσω του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το κοινό πρόγραμμα. Ε, έχει φτάσει το μήνυμα της προσπάθειάς μας για τη δημιουργία αυτού του κοινού προγράμματος στις φαρμακευτικές εταιρείες και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή μαζί τους διότι οι έρευνες οι οποίες γίνονται από τις εταιρείες αυτές είναι πανάκριβες και αναγκαίες. Επειδή λοιπόν χρειάζεται ε, ένα ουσιαστική χρηματοδότηση πρέπει να, σαφώς να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και ε, να συντονίσουμε τις ερευνητικέ προσπάθειες που γίνονται στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το κοινό πρόγραμμα. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη προαιρετικά, εθελουσίως, ε, να συμμετάσχουν σε αυτό το κοινό πρόγραμμα. Δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες δομές. Από ό,τι έχουμε ε, κατανοήσει από τα κράτη-μέλη, ε, μπορούμε να συντονίσουμε ένα δίκτυο επιστημονικών συμβούλων, ε, ερευνητικών κέντρων και έτσι μπορούμε σαφέστερα να εντοπίσουμε τι χρειάζεται να επιτύχουμε, τι θέλουν τα κράτη-μέλη, τι επιδιώκουν, τι θέλουν να κάνουν, να καταφέρουν για να μπορέσουν να συντονίσουν καλύτερα τα ερευνητικά τους προγράμματα. Τώρα, ρωτήσατε ποιος ε, είναι ο ρόλος της Κομισιόν ε, σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε facilitators, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο είμαστε ο σύνδεσμος, είμαστε το όργανο το οποίο διευκολύνει και συντονίζει ε, όλη αυτή την προσπάθεια ε, θα εντοπίσουμε πού υπάρχουν τα κενά και οι ελλείψεις ε, για να διοχετεύσουμε τις πληροφορίες αυτές στα κράτη-μέλη, να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε λοιπόν ε, όλες τις πτυχές που χρειάζονται για την ανάπτυξη της έρευνας. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα γεμίσουν τα κενά και θα συμπληρώσουν συνολικά την εικόνα ε, ώστε να είναι πλήρης για να μπορέσουμε ακριβώς να ολοκληρώσουμε αυτό το συντονιστικό πλαίσιο. Βέβαια είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για την κοινωνία και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στην πρόληψη. Πρέπει να ε, κατανοήσει, πρέπει να αυξήσουμε την, την γνώση, την κατανόηση του Ευρωπαϊκού, των Ευρωπαίων πολιτών στις ασθένειες αυτές. Ε, το γεγονός είναι ότι είναι μια προτεραιότητα στην έρευνα είναι αυτές οι ασθένειες. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να, αυξήσουμε την ενημέρωση των πολιτών και σε αυτές τις ασθένειες ειδικά, αλλά και σε όλα τα θέματα υγείας. Διότι όπως λέγανε και οι αρχαίοι νους υγιείς εν σώμα τη All um, uh, Εάν λοιπόν εξετα... Ε, μελετήσετε την ε, έρευνα η οποία εμπλέκεται σε αυτό τον τομέα ε, θα διαπιστώσετε ότι είναι ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρούς ουσιαστικούς επιστήμονες που δεσμεύονται σε αυτό το θέμα και σαφώς προσπάθειά μας είναι να προσελκύσουμε τα καλύτερα μυαλά για να μπορέσουν να εξετάσουν ε, και να αναπτύξουν την έρευνα και ε, σε όλες τις υπήρους βεβαίως θα καλύψει αυτό ο συντονισμός μας. Ε, θα μελετούμε και τις ε, καρδιογγειακές ε, ασθένειες, τις, το διαβήτη, τις προκύπτουσες επιδημίες, όλα αυτά βεβαίως. Μια πλήρης ενημέρωση όλων των θεμάτων υγείας παγκοσμίω υπάρχει σε μας και τις έχουμε κατά νου. better Ένας από τους βασικούς στόχους μας όπως ε, ρωτήσατε είναι η εστίαση ε, που, που, ακριβώς συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και θα διαθέσουμε τα χρήματά μας ε, για να μην γίνονται ανώφελες πατάλες. Σύμφωνα με τις στατιστικές θα διπλασιαστεί ο ρυθμό των πασχόντων από Alzheimer σε 10-15 χρόνια και το σε, 50, σε 40 χρόνια, όπω είπαμε, το 2050 θα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν μια τεράστια πρόκληση αυτή. I hope that I've addressed all your... <laughs> Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας συνοπτικά και εάν θέλετε μπορείτε να μου τις ε, υποβάλλετε γραπτό ή να μου στείλετε ένα μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας απαντήσω. Θα είμαι ευτυχής να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων πάρα πολύ θερμά. Σας ευχαριστώ για τις τόσο εκτενείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σας. Μα κεντρήσατε ίσω λίγο περισσότερο την περιέργεια για αυτό το σημαντικό θέμα και αυτό είναι ακριβώ το σημαντικότερο που πετύχαμε σήμερα γιατί είναι προπόθεση για να προχωρήσουμε και να σας στηρίξουμε κι εμείς πολύ για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ, ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα και ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το σημείο σημείο διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα και μετά πάμε στις ψηφοφορίες, έτσι. Ένα λεπτό, μισό λεπτό, ό,τι θέλετε να βγάλετε τις κάρτες και να ετοιμαστείτε. Για να φτάσουν και οι τελευταίοι συνάδελφοι. Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε όλοι παρόντες, απάντηση ναι. Έχετε τις κάρτες σας. Έχετε την κάρτα ψηφοφορία σας, δεν θα ψηφίσουμε. Κυρίες και κύριοι, θα επιθυμούσα να αρχίσουμε τώρα ψηφοφορίες. Ή να συνεχίσουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Έχουμε και τις κάρτες ψηφοφορίας μας όλοι και η δική μου είναι εδώ και δουλεύει ελπίζω. Sie Also, meine Damen Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πρώτο σημείο είναι η ψηφοφορία για την απλοποιημένη διαδικασία 46.1 Διεθνής ε, Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ρένα. Εδώ πρέπει να πούμε ναι ή όχι μόνο. Και έχω αναλάβει αυτό το σημαντικό έργο να παρουσιάσω όλη την τεκμηρίωση ή μάλλον η γραμματεία μας έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα ε, για να προσθέσουμε ή όχι αυτή την πρόταση. Μπορώ να υποθέσω ότι όλοι συμφωνείτε με την προσθήκη. Αντιρρήσεις, καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία, συμφωνούμε σε ε, ε, αντίρρηση ο κύριος... Όχι, όχι. Υπέρ, υπέρ. Α, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ότι Εγκρίναμε αυτή την τροπολογία. Ε, η κυρία ΕΚ για τον προϋπολογισμό ως εισηγήτρια μας υπέβαλε μια πρόταση. Υποθέτω ότι έχετε όλοι όλο τον κατάλογο ψηφοφορίας. Λοιπόν, αρχίζουμε. Καταρχάς, τροπολογία 1, υπέρ, υπέρ. Ε, κατά. Εγκρίνεται 2, 2, τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τρία. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, μερικές ψήφοι κατά, αλλά ε, υπερψηφίζεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, είμαστε σίγουροι. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένουμε λίγο την Αντιπρόεδρο, ωραία. Έληξε ψηφοφορία. Όχι. Ποιο δεν έχει κάρτα. Δεν, δουλεύει κάρτα. Ο, ο κύριος Γκλάντε. Α, δεν έχει πάρει ακόμα την καινούργια κάρτα του. Πέστε μου σας παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος, ε, ε, ποιος έχει πρόβλημα, δείξτε μου. Ποιος έχει πρόβλημα. Ποιος έχει πρόβλημα με την κάρτα παρακαλώ. Ψηφίζουμε λοιπόν καταρχάς και μετά ε, χειρό χειρός θα ψηφίσουμε αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, έληξε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα είναι Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω αυτού που έχουν ελαττωματική κάρτα να ψηφίσουν. Ποιο είναι υπέρ, υπέρ. Κανεί κατά, τρι, τε, πέντε, πέντε. Άρα λοιπόν έχουμε. οι 12 υπέρ και 32 κατά, τρει αποχές. Σωστό, έξοχα. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε όλο το πακέτο. Ποιο συμφωνεί, ποιο υπερψηφίζει. Κατά. Α, ηλεκτρονικά. Ας το κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα. Έληξε, έληξε η ψηφοφορία να ψηφίσουν τώρα αυτοί που δεν, έχουν τις, δεν είναι εντάξει οι κάρτες τους. Ποιος παρακαλώ ψηφίζει υπέρ. Α, λειτουργήσαν οι κάρτες σωστά. Έχουμε 43 υπέρ, 6 αποχές. Ε, υπέρ ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, πολύ ωραία. Άλλα σχόλια παρατηρήσεις για την ψηφοφορία, όχι. Και έτσι προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι η επίσκεψη της κυρίας Επιτρόπου η οποία δεν είναι ακόμα εδώ αλλά δεν μπορεί να μας επισκεφθεί ε, πρέπει να περιμένουμε να περιμένουμε λιγάκι αγαπητοί συνάδελφοι έχετε το νου σας μόλις έρθει θα ξεκινήσουμε δεν θα κάνουμε μεγάλο διάλειμμα Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße in ihrer aller Καλωσορίζω εξ ονόματος όλων την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ για πολλωστή φορά στην Επιτροπή μας και έχουμε την ευκαιρία μαζί της να συζητήσουμε θέματα της αρμοδιότητάς της και θα οργανώσουμε τη συζήτηση ως εξής. Η κυρία Επίτροπος θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση καταρχάς για να έχουμε μια βάση συζητήσεως και με... μετά θα πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά ε, και με ενδιαφέρον. Δίνω το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω το καλύτερο είναι να μιλήσω αγγλικά, γιατί περισσότεροι θα με καταλάβουν έτσι παρά να μιλήσω λουξεμβουριανά. The um, Ας έρθουμε στην ουσία. Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία 2010 προκειμένου να ελέγξουμε κατά κάποιο τρόπο την οικονομία της ενιαίας αγοράς για τα ψηφιακά και να βελτιώσουμε τη θέση της έρευνας της ICT για έρευνα και καινοτομία και όλα τα ωφέλη να είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες. Σημειώθηκε πρόοδος σε αυτή την ενιαία ψηφιακή αγορά γιατί καταφέραμε να ε, ομαδοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και τα οπτικοακουστικά. Και δεν χρειάζεται να σας θυμίσω την, το τι ήταν επιτυχία οι κανονισμοί για το roaming, την περιαγωγή του 2007-2009. Και έτσι από κοινό αντιμετωπίσαμε μια αποτυχία της ενίας αγοράς με συγκεκριμένα ωφέλη για όλους τους Ευρωπαίους χάρη σε μια ομαλή λειτουργία διαδικασία συναπόφασης ε, οργανώσαμε τη συμφωνία αυτή σε χρόνο ρεκόρ. Γενικά <clears throat> οι Ευρωπαίοι πολίτες εποφελούνται από τις φτηνές τιμές και τη σταθερή τηλεφωνία. Είχαμε μείωση 27% τα τελευταία χρόνια, σε τέσσερα τελευταία χρόνια των τιμών. Συχνά δεν το αναφέρουμε αυτό. Το κόστος για τα κινητά πέραν της περιαγωγής μειώθηκε κατά 34% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Για την περιαγωγή, το roaming, όπως ξέρετε, οι τιμές μειώθηκαν κατά 70% από το 2005. Θα συνεργαστούμε επίσης στο θέμα αυτό και στο μέλλον. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια ενδιάμεση έκθεση του χρόνου και η πλήρη αναθεώρηση ανασκόπηση μάλλον το 2011. Εκεί στην πλήρη αυτή ανασκόπηση θα εξελογήσουμε όλες τις εξελίξεις στην αγορά και στην τεχνολογία. Επίσης η Επιτροπή σας βόηθησε στο να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο για τις δορυφορικές υπηρεσίες, το περίφημο FSS, σε λιγότερο από 10 μήνες. Μια ενιαία διαδικασία για επιλογή φορέων για τις δορυφορικές επικοινωνίες ήδη υπάρχει από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η έγκριση σε εθνικό επίπεδο, οι δύο επιλεγμένοι φορείς, η Μερσάτ και Solaris, θα αναπτύξουν το σύστημα αυτό κινητής τηλεφωνίας δορυφορικά το αργότερο μέχρι το 2011 και η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης αυτής, όπως το θέλησε και το Κοινοβούλιο και αυτό θα καλύπτει όλη την έκταση, τη γεωγραφική έκταση της Ένωσης. Έρευνα. Για να μειωθεί ένα κενό που έχουμε στην τεχνολογική έρευνα, στη σύγκριση με άλλες οικονομίες στον κόσμο, δώσαμε τον πιο μεγάλο προπολογισμό για την έρευνα ICT μέχρι τώρα, πάνω από 10 δις ευρώ, 2007 μέχρι 2013. Αυτή η χρηματοδοτούμενη έρευνα της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιομηχανία. Τονίζω την επιτυχία στην νάνο ηλεκτρονική, μικροηλεκτρονική, στην ασφάλεια, στην οδική, στις οδικές μεταφορές, όπου η έρευνα πέρασε άμεσα, άμεσα, αμεσότερα σε βιομηχανικές εφαρμογές. Επίσης, έχουμε το νέο σύστημα κοινής, ε, πρωτοβουλειών κοινής τεχνολογίας, μια εταιρική σχέση δηλαδή ιδιωτικού και δημόσιο τομέα. Όπως ξέρετε έχουμε, έχουμε δύο τέτοια προγράμματα νανοτεχνολογία και embedded systems όπως τα λέμε. Βέβαια εδώ είμαι κάπως απογοητευμένη από τα κράτη-μέλη διότι θα μπορούσαμε να, θα να είχαμε δαπανίσει 25% περισσότερο αν οι χώρες μέλη έδιναν τα λεφτά που είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν. Επιμένω λοιπόν ο κάθε εταίρος, το κάθε μέρος της συμφωνίας αυτής να παίξει πλήρως το ρόλο του. Άλλη κοινή δράση, ένα πρόγραμμα ε, για το πώς να γερνάμε καλύτερα, έτσι το λέμε στη βιομηχανική μας κοινωνία. Εδώ τρεις χώρες παίρνουν μέρος. Μιλάμε για 600 εκατομμύρια 2008 έως 2013 με πολύ συγκεκριμένους στόχους στην έρευνα για τους ηλικιωμένους και άτομα που έχουν ε, προβλήματα προκειμένου να προσαρμοστούν σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, με βοήθεια νέων τεχνολογιών. Εδώ έχουμε 40 πανευρωπαϊκά προγράμματα προς χρηματοδότηση και τα κράτη-μέλη αύξησαν την αρχική συνεπένδυση κατά 40%. Στον τομέα αυτό δηλαδή τα πάνε καλά τα κράτη-μέλη και η σημαντική μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στο 43%. Στο 43%. Σας προλαβαίνω για τις ερωτήσεις που θα κάνετε. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργότατα. Περαιτέρω πρόεδρο μετά από μερικούς μήνες θα σας κάνω αναφορά. Ποιότητα ζωής και μη αποκλεισμό. Ένα πολύ σημαντικό για την μερίσια διάταξη του Κοινοβουλίου σε κοινή δήλωση δηλώσαμε στις 11 Φεβρουαρίου ημέρα 112 ημέρα 112 προκειμένου να προωθεί αυτό το 112 Μπορεί κανείς να τηλεφωνήσει και από σταθερό τηλέφωνο και από κινητό το 112 σε όλες τις χώρες μέλη. Μεγάλη πρόοδος αυτή. Γιατί όταν ξεκινήσαμε το 112 πριν από 5 χρόνια, στην αρχή δεν έπαιρναν πολύ αυτό το νούμερο. Βέβαια έχουμε ακόμα μερικά προβλήματα σε μερικές χώρες μέλη ε, το παρακολουθούμε από κοντά το πρόβλημα προκειμένου να το επιλύσουμε. Τι μάχες δίνουμε αυτή τη στιγμή. Θυμόστε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στην Επιτροπή σας, για τη μελλοντική χρήση του ψηφιακού μερίσματος. Αυτό ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, με την έκθεση Τόγια καλό παράδειγμα συνεργασίας Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πολιτική και κοινωνικονομική διάσταση ενός ερωτήματος που όλοι στην αρχή θεωρούσαμε τεχνολογικό πρόβλημα ή ερώτημα. Ε, δεν είναι μόνο τεχνολογικό, έχει επίπτωση και, στην, και στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται όταν η αναλογική τηλεόραση θα αλλάξει. Ξέρετε έχουμε ορίσει την χρονολογία στο 2012 για την αλλαγή αυτού του είδους της τηλεόρασης. Οι ευκαιρίες αυτές αφορά και το ευρύ φάσμα αλλά και άλλους τομείς προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση ευρέως φάσματος και σε άλλες, για άλλες υπηρεσίες προκειμένου να ξεπεράσουμε το ψηφιακό χάσμα. Μετά από την προπαρασκευαστική δουλειά, μετά από πολύ σοβαρή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, Κάποια στιγμή θα είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω μία ανακοίνωση. Αυτό θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, στους επόμενους μήνες, εσείς κύριε Πρόεδρε, θα έχετε το κείμενο αυτό μπροστά σας. Επίσης, θα συζητηθεί επίπεδευτή σε στρατηγικό επίπεδο με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με στα πλαίσια της του πρώτου προγράμματος στρατηγικής για το φάσμα, προκειμένου να ορίσουμε μέτρα που είναι αναγκαία προς έγκριση με συναπόφαση. Και ελπίζουμε αυτή η συζήτηση να ξεκινήσει στην διάσκεψη για το φάσμα που θα την οργανώσει το Κοινοβούλιο. Από ό,τι ξέρω, θέλετε τη διάσκεψη αυτή για το σπέκτρουμ, για το φάσμα, την κάνετε τον Ιανουάριο. Εν πάση περιπτώσει, η Κομισιόν θα έχει κάνει την προπαρασκευαστική δουλειά μέχρι τότε προκειμένου η διάσκεψη αυτή κορυφή σας την πούμε να είναι επιτυχής. Κοινός μας στόχος είναι μια, ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον και ένα κοινό όραμα για καλύτερες υπηρεσίες και πρέπει να αναθεωρούμε την πολιτική μας περιοδικά για να προσαρμοζόμαστε στην εξελισσόμενη κατάσταση. Από κοινού. ίντερνετ με ευρύ φάσμα. Ξέρετε, είναι ζωτική σημασία για το πρόγραμμα ανάκαμψη Γι' αυτό έχουμε βρει περίπου ένα δις εκό προκειμένου να ε, καλυφθούν και χώροι της υπαίθρου με την ευρυζωνική αυτή χρήση του ίντερνετ, του διαδικτύου. 30% αυτών που ζουν στην Ήπεθρο δεν έχουν πρόσβαση καθόλου σε ευρυζωνικό διαδίκτυο. Είμαι απογοητευμένη και γι' αυτό. Για το ότι μερικές χώρες ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να επωφεληθούν από τα νέα αυτά κονδύλια για τα προγράμματα ανάπτυξη τη υπαίθρου που μας έχουν υποβάλει. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε μαζί τους γιατί πρέπει να σπάσει αυτό το φράγμα, αυτό το ψηφιακό χάσμα. Είναι ευθύνη όλων των πολιτικών αυτό. Αυτή είναι η τρέχουσα δουλειά. Τώρα περνάω στο τι χρειάζεται να κάνουμε στο άμεσο μέλλον για να πετύχουμε τις προτεραιότητές μας. Όπως ξέρετε, σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές επενδύσεις και την οικονομία και ο πρόεδρος Βαρόσο το είπε σαφώς στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η επόμενη Κομισιόν θα περάσει, από μια ψηφιακή, θα περάσει σε μια ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να συνδέεται με τα διαδίκτυα του μέλλοντος. Θέλουμε να έχουμε ευρυζωνικό διαδίκτυο για τους 27 και εδώ τίθεται το θέμα του ψηφιακού χάσματος και το τι επενδύσεις απαιτούνται για να καλυφθεί και αυτό το 30% της του χώρου που δεν καλύπτεται σήμερα και το 2013 ε, ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας για όλους. Αυτή είναι οι δύο στόχοι. Για να έχουμε ανταγωνιστική υποδομή για μια ψηφιακή Ευρώπη απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για τους επόμενους μήνες μάλιστα. Γνωστά αυτά. Ανταγωνισμός, βιώσιμη ανάπτυξη στα διαδίκτυα νέας γενιάς πρέπει να περάσουμε στις ίνες. Και όταν λέω νέας γενιάς δεν λέω να κάνουμε αναβάθμιση με χαλκό, οπτικές ίνες. Δεύτερο, η υπηρεσία των κινητών πρέπει να είναι πιο ελκυστική και να στρώσουμε κατά κάποιο το δρόμο για τη νέα γενιά κινητών. Ε, προηγούμαστε στα κινητά σε σχέση με άλλες υπήρους δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Γι' αυτό πρέπει να περάσουμε από το 3G στο 4G. Και τέλος, το πέρασμα από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση πρέπει να επιταχυνθεί. Γιατί αυτό θα απελευθερώσει μεγάλα κομμάτια φάσματος που σήμερα χρησιμοποιείται από ε, αναλογική τηλεόραση εδάφους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα από νέες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία δηλαδή εδώ, ας την εκμεταλλευτούμε. Δεδομένης της υποδομής, Γίνεται το πρόβλημα. Όχι βέβαια, διότι το, το διαδίκτυο απαιτεί ελκυστικές υπηρεσίες για όλους τους χρήστες και πολλές επαφές πέραν φύλου, κοινωνικής κατάστασης κλπ. Γι' αυτό η Κομισιόν ξεκίνησε μια ευρεία διαβούλευση για τις προτεραιότητες για μελλοντικές πολιτικές. Αυτή η διαβούλευση θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου μάλλον, και μετά θα έχουμε μια διάσκεψη. Από ό,τι ξέρω κύριε Πρόεδρε, μερικά μέλη της Επιτροπής σας θα πάρουν μέρος. Μέχρι στιγμής με την ευρύ αυτή δημόσια διαβούλευση είχαμε 410 απαντήσεις, πολύ υψηλού επίπεδου, 85% αυτών των απαντήσεων προέρχονται από ιδιώτες. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Σημαίνει ότι σιγά σιγά περνάμε στο επίπεδο του πολίτη. Πέραν των προκλήσεων που ανάφερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τέσσερις άλλες προτεραιότητες. Προσδράση για να έχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά. με τους χρήστες του διαδικτύου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέτουν ερωτήματα σχετικά με το δικαιώματα του καταναλωτή και το ίντερνετ, ελευθερία παροχής υπηρεσιών online διασυνοριακά και δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι καταναλωτές στο διαδίκτυο. Πολλές φορές διαπιστώνουν ότι εκεί που ζουν δεν έχουν πρόσβαση σε εμπορικέ υπηρεσίες σε σχέση με οπτικοακουστικό περιεχόμενο που θα μπορούσαν να έχουν στο σπίτι τους πέραν των συνόρων. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Η πρώτη προτεραιότητα. Να το κάνουμε αυτό πιο, να το διευκολύνουμε. Το, την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο οπουδήποτε παράγεται στην Ευρώπη. Το να υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο ελκυστικό για τους πολίτες μας θα είναι αποφασιστικό προκειμένου να προωθηθεί το ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλή ταχύτητα. Δεν αρκεί δηλαδή η υπόδομη. Χρειαζόμαστε και μια πολιτική υπηρεσιών και περιεχομένου ταυτόχρονα. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς. Δεύτερη προτεραιότητα. Ασφαλές, ασφαλής χώρος και φιλικός προς το χρήστη όσον αφορά τις πληρωμές για τα κινητά. Σήμερα δεν υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές για το ΆΜΚΑΣ με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλευόμαστε όλο το δυναμικό που υπάρχει. Έχουμε περισσότερους από 500 εκατομμύρια χρήστες κινητών στην Ευρώπη. Αν τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν τα κινητά τους για κάθε είδους εφαρμογή, ο κλάδος αυτός θα γίνει πολύ πιο ισχυρός. Τρίτη προτεραιότητα, άνοιγμα προς τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουμε 23 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 23 εκατομμύρια, το 99% όλων των επιχειρήσεων. 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά στη χρήση της προκειμένου να προωθεί η παραγωγικότητα μέσω αυτών που συζητάμε, καθυστερούμε, καθυστερούμε σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, μόνο το 9% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ε, ηλεκτρονική τιμολόγηση. 11% ε, ε, ε, χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές για τους ανθρώπινους πόρους. Αν είχαν καλύτερη πρόσβαση και μέσω του Ιντερνετ με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν, δεν θα χρειαζόταν να αγοράζουν άλλου είδους υπηρεσίες. Το cloud computing, που είναι ένα, κάτι το κενό, με θετικά και αρνητικά, θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να υποφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν το καταφέρουμε, πώς θα, μπορέσουμε να αποφύγουμε τις τυχόν παγίδες. Τέταρτη προτεραιότητα, καλύτερη χρήση καινοτομιών σε σχέση με την ηλεκτρονική τεχνολογία. Την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν θα ε, δημοσιεύσει μία σύσταση για το ICT και την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας πράσινο ICT. Νομίζω είναι μια από τις μελλοντικέ εξελίξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και για τη βιομηχανία γενικότερα προκειμένου να έχουμε νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας. Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα που ανάφερα, η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ψηφιακή στο σύνολό τη με μια νέα στρατηγική της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλους τους χώρους της πολιτικής. Ο πρόεδρος της Κομισιόν σας πρότεινε να συσταθεί μια ψηφιακή οικονομία. Η Επιτροπή σας καλείται να κάνει αυτή τη δουλειά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την εμπεριστατωμένη αυτή η παρουσίαση προγραμμάτων τα οποία αναπτύσσονται, τα οποία, με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε άμεσα και πιστεύω ότι έχουμε μία θαυμάσια βάση συζητήσεως. Ε, η κυρία Τράουτμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για αυτή την επισκόπηση που μας ε, κάνατε. Διαπιστώνω ότι δεν καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, έθεσε σε ισχύ ε, όσα είχε αναλάβει για την πολιτική του φάσματος και το δικό χάρτη όπως είχε ονομαστεί και χαίρομαι που ήδη συμπεριλαμβάνεται το Κοινοβούλιο στην προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής που ελπίζω όπως και εσείς να γίνει το Ιανουάριο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να δούμε τι θα κάνουμε για το ραδιοφάσμα στο μέλλον. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις τώρα για θέματα τα οποία δεν θίξατε ιδιαίτερα. Ε, θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω ε, πώς βλέπετε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης που το είχατε παρουσιάσει ως προτεραιότητα, αλλά τελικά στις επόμενες προτεραιότητες δεν συμπεριλαμβάνεται. Είναι επίκαιρο το θέμα και στην ίδια μου τη χώρα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς σε σχέση με αυτό, ε, τι γίνεται με την online ε, έκδοση. Σήμερα ανησυχούν πάρα πολύ επιστημονικές και δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη γιατί υπάρχει μία συγκέντρωση σε τέσσερους, ε, τέσσερους εκδοτικούς οίκους επιστημονικούς σε όλους τους κλάδους και ένα θέμα είναι η αρχιοθέτηση των πηγών που κανονικά ε, πληρώνει κανείς και για να έχει πρόσβαση στις βιβλιοθήκες αλλά αν σταματήσει αυτό το εγχείρημα θα σταματήσει και η πρόσβαση. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Πληρώνουν οι βιβλιοθήκες για να έχουν πρόσβαση και για τη διάρκεια δεν έχουν καμία εγγύηση για τις πηγές αυτές, τις οποίες έχουν πληρώσει όμως. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί, πιστεύω. Θα ήθελα επίση να σα ρωτήσω για το πρόβλημα των προτύπων και προδιαγραφών. Σήμερα έχουμε πολλέ εταιρείε, ιδιαίτερα ε, μικρομεσαίε και startup που ασχολούνται με την παραγωγή νέου περιεχομένου και νέων υπηρεσιών. Τι ε, ε, τίθεται λοιπόν το ερώτημα τη στρατηγική που μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρότυπα και προδιαγραφέ. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Και μια τελευταία ερώτηση και σημαντικό πάλι το θέμα που αφορά το περιεχόμενο και τη πνευματική ιδιοκτησία. Εμείς ε, ξεκινήσαμε σε μια ομάδα εργασίας, μια δουλειά, ο προείδρευε ο κύριος Τουμπό και εκπροσωπεί το και η δική μας επιτροπή και ήθελα να μάθω και πάλι στην προοπτική του περιεχομένου στο διαδίκτυο που είπατε ότι είναι και προτεραιότητα. Σήμερα τι λέτε Πώς θα χειριστείτε αυτό το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και το cloud computing και ε, την εξέλιξη της χρήσης του διαδικτύου, η οικονομία της γνώσης είναι εφικτή εάν δεν αποφανθούμε για την ουδετερότητα του δικτύου. Τέσσερις ερωτήσει σας έκανα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν σημαντικές όμως και τέσσερις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αγαπητή Βιβιάν για αυτή την παρουσίασή σου. Ε, καταρχάς σας ε, ε, συγχαίρω για το, πρόγραμμα υποβοηθούμενης ε, διαβίωσης ή μάλλον ναι, της ε, καλής γύρανσης. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δημογραφικά γυράσκουμε και είναι μια ήπειρος όπου αυξάνονται ηλικιωμένοι, και πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Είναι σωστό να συμπεριλάβουμε και αυτό το θέμα της αξιοπρεπούς γύρανσης μαζί με το Alzheimer επειδή ακριβώς εμείς ως Ευρωπαίοι μας θίγει ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό της γύρανσης, της μακροβιότητας του πληθυσμού. Τώρα, πώς θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα αυτό επειδή η χρηματοδότηση είναι πολύ πτωχή. Γι' αυτό χρειάζεται μια συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου ε, και Συμβουλίου ε, και Κομισιόν για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερα τη χρηματοδότηση αυτού, αυτών των προγραμμάτων και οτιδήποτε αφορά τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων θα το υποστηρίξουμε. Όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και το copyright, Θέλω να παρατηρήσω το εξή. Όλο και περισσότεροι τομεί τη βιομηχανία μα ή τη οικονομία μα, συγγνώμη, ε, οδηγούνται προ το ίντερνετ. Αλλά προκύπτουν συνεχώ προβλήματα προστασία ε, δεδομένων και πνευματική ιδιοκτησία. Είναι λοιπόν ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρο. Εμεί δεν είμαστε αυτό το οποίο οι οποίοι τα επιτρέπουμε όλα, ελευθερία, ελεύθερη χρήση σε όλα όπω οι Αμερικανοί ή καμία ελευθερία ε, για το ίντερνετ όπω οι Κινέζοι. Κάπου πρέπει να βρούμε ε, τη μέση οδό, τη χρυσή τομή. Πολλά προβλήματα έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, πολλά ερωτήματα έχουν ε, ανακύψει και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν εάν το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου μπορεί να συμπληρωθεί και με το θέμα της προστασίας της ασφάλειας δεδομένων. Εκεί δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην ιδανική κατάσταση όπου όλα τα δεδομένα προστασία δεδομένων ε, ε, είναι εξασφαλισμένη και στεγανή. Ε, Επίση, οι αξιόπιστες πηγές, η χρήση των αξιόπιστων πηγών. Ποιε είναι αυτέ αυτές οι trusted sources. Μιλάμε πάντοτε για το περιεχόμενο και το περιεχόμενο. Το πρόβλημα όμως είναι ποιε είναι οι πηγές, από πού προέρχεται αυτό το περιεχόμενο. Διότι έχουμε μία ε, χιονοστιβάδα περιεχομένου η οποία μας καταπλακώνει αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πηγές από πού προέρχονται όλα αυτά τα δεδομένα και αν είναι αξιόπιστες. Ποιοι είναι οργανισμοί, τα ιδρύματα τα οποία είναι πιστοποιημένα και, από τα οποία, και στα οποία μπορούμε να βασιστούμε ότι έχουν τις αξιόπιστες πηγές. Είναι μια διαδικασία την οποία έχετε ξεκινήσει και πιστεύω ότι χρειάζεται να ολοκληρωθεί συνεχεία την ευρυζωνική, η προσπάθεια για ευρυζωνική, ε, η ευρυζωνικό διαδίκτυο, ευρυζωνική σύνδεση. Το υποστηρίζω πλήρως. Εκεί όμως που ακόμα έχουμε λήψει είναι ο συντονισμό της δικής σα πρωτοβουλίας με την, το συντονισμό των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της υπαίθρου, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ξέρω ε, ότι εσείς ιδιαίτερα έχετε ασχοληθεί και έχετε συζητήσει τα θέματα αυτά με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, το ξέρω αυτό. Και τώρα που ε, ε, επανακαθορίζουμε την περιφερειακή πολιτική πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε αυτό το θέμα, ειδικά το συντονισμό της, ε, των πολιτικών, την ανάπτυξη της αποτολισματικότητας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ρεύμα από την Κομισιόν, ένα ρεύμα συνεργασίας για να συνδυάσουμε το ευρυζωνικό θέμα με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ευχαριστώ. η κυρία Νταλκαστίγιο. Eh, Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, για την παρουσία σας σήμερα εδώ, αλλά και την παρουσίασή σας. μας παρουσιάσετε συνοπτικά ε, το που βρισκόμαστε και κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά όλα εκτενέστερα όταν θα γίνουν οι ακροάσεις των επιτρόπων, των υποψηφίων επιτρόπων. Πάντως και σήμερα είναι καλή ευκαιρία γιατί μέχρι τώρα εσείς ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα που συνδέονται μεταξύ τους και ένα τρίτο που είναι ένα θέμα ακόμα και πάντα σε εκκρεμότητα. Θα σας το πω μετά. Τα δύο πρώτα που συνδέονται μεταξύ τους είναι αφενός αυτό που έχει να κάνει με το ραδιοφάσμα, το ψηφιακό χάσμα, τη ε, μετάβαση από την αναλογική πραγματικότητα στην ψηφιακή και την ευρυζωνικότητα. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, διότι η δυνατότητα πρόσβασης ασφαλούς και ταχεία στο διαδίκτυο είναι κάτι που ευνοείται πάρα πολύ από τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ε, κανείς ε, κάποια ε, μέρη του φάσματος που θα απελευθερωθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Η πολιτική εκεί, διάφορα κράτη-μέλη διαφέρει ανάλογα με το ραδιοφάσμα ανάλογα αν τα κράτη διαχειρίζονται αυτά τα θέματα με τρόπο που να συνεισφέρει και να υπάρχει μια ανάπτυξη έτσι πιο ταχεία των ηλεκτρονικών ε, επικοινωνιών με μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα. Από την άλλη υπάρχουν κάποιες χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επικοινωνία με άλλο τρόπο, παραμένει αναλογική η τηλεόραση και θα υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ότι είναι άμεση η προτεραιότητα. Θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα εξισορρόπησης. Αυτό το ραδιοφάσμα που θα απελευθερωθεί είναι πολύ καλό για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες. Δεύτερον, η ανάπτυξη αυτή της ψηφιακής Ευρώπης που αναφέρατε. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το να υπάρχει και μια λεωφόρος, μια δόση ανάπτυξης, εντάξει, διαδίκτυο, ευρυζωνικότητα κτλ. Αλλά εκτός από αυτό έχει πολύ μεγάλη σχέση με το να είναι εξοικειωμένο ο κόσμος, να ξέρει να χρησιμοποιεί, να έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ. Δηλαδή, και σε πολλού τομεί από το ηλεκτρονικό εμπόριο και πολύ διαφορετικού. στη δημόσια υγεία ή ε, στην εκπαίδευση ή στην ενέργεια. Ε, έχει πολλές εφαρμογές. Όλοι αυτοί οι τομείς λοιπόν για διάφορους λόγους χρειάζεται ο κόσμος να χρησιμοποιεί άμεσα αυτό το εργαλείο. Μπορεί λοιπόν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, δραστηριότητες καθημερινής ζωής να περάσουν από το διαδίκτυο και αυτό είναι και πολύ αποτελεσματικό και πολύ αποδοτικό. Αυτό είναι το σύστημα. Αλλιώς την ευρυζωνικότητα γενικά τι να την κάνω στην Ήπεθρο. Καλό είναι, μου αρέσει, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί ο κόσμος να το χρησιμοποιεί. Ή έστω και υποχρεωτικά να ε, συνδιαλέγεται ο κόσμος με τις ε, υπηρεσίες υγείας, παιδείας έστω και το εμπόριο στην καθημερινή του επαναλαμβάνω ζωή. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή έχουν πολύ μεγάλο νόημα όλες οι τομεακές και κλαδικές πρωτοβουλίες αν θέλουμε πραγματικά την ψηφιακή Ευρώπη. Και ένα τρίτο, μέγα ζήτημα που εκκρεμεί καιρό και είναι και επίμαχο θέμα. Το copyright και τα περίφημα πνευματικά δικαιώματα, η πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό είναι θέμα που κανένας δεν έχει λύσει υπάρχει ακόμα και εκρεμεί και ε, προκαλεί πολλά προβλήματα κάθε είδους σε όλες τις χώρες. Αυτή θα πρέπει λοιπόν να είναι η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να προσπαθήσουμε να λύσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα και να απαντήσουμε σε αυτή την ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φων Μίσλχοφ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε δύο ε, παρατηρήσεις. Μας ενημερώσατε για τις δραστηριότητες ε, που ξεκινήσατε για τις καινοτομίες για την ηλεκτρονική πραγματικότητα και των επιχειρήσεων που θα πρέπει να επενδύσουν και οι εταιρείε για την έρευνα και την ανάπτυξη. Τώρα μας λέτε ότι υπάρχουν δισταγμοί στην εκτέλεση και παραπέμπεται στα κράτη-μέλη. Αυτό έχει να κάνει με την κρίση, ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέσα οικονομικά ή υπάρχει κανένα λάθος στην ε, κατασκευή του όλου εγχειρήματο, πώς να το ε, στην ατζέντα και στην εφαρμογή, αν θέλουμε να βοηθήσουμε. Μπορεί να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά δεν θα πρέπει να πιέζουμε. Ξέρουμε ότι ζούμε έκτακτους καιρούς, αλλά αυτοί οι καιροί θέλουν και έκτακτες λύσεις και για την υποστήριξη πραγματικά στην καθημερινή ζωή είναι μικρός ο προπολογισμό τελικά μου φαίνεται. Αν ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα στα κράτη-μέλη, ίσως θα πρέπει από κοινού να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, γιατί αυτό γίνεται και, και, και μπορούμε να το κάνουμε. Είναι καλή εξέλιξη θετική. Ξέρω ότι προσεχώς το Κοινοβούλιο θα συζητήσει αυτό το θέμα με όλους τους εκπροσώπους των ηλικιωμένων στην Ευρώπη διοργανώνουμε μία διάσκεψη για να τους ε, ενημερώσουμε για αυτή την ευχάριστη είδηση. Καλά όλα αυτά. Και ρωτώ τι κάνετε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση συγκεκριμένα. Ευχαριστώ συνάδελφα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω δύο θέματα να θίξω. Καταρχάς το ICAN. Η σύμβαση αυτή λύγει στις 39 του με το ε, ε, αντίστοιχο Υπουργείο των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρατε τις, υποδομέ υποδομές και όλο το, την, την κατεύθυνση που θέλουμε να λάβει το ίντερνετ. Όλα αυτά τώρα ε, εξαρτώνται από το ICAN και έναν κυβερνητικό, μη κυβερνητικό οργανισμό και θα ήθελα να ξέρω πώς θα συνεχίσετε την εξέλιξη του ICAN μετά τις 30 Σεπτεμβρίου με τους Αμερικανούς και το Υπουργείο Εμπορίου. Εν συνεχεία, το πακέτο τηλεπικοινωνιών θα με ενδιέφερε πώς η Κομισιόν ε, τι θέση έχει η Κομισιόν στο θέμα της ε, του διαδικτύου και τι θέση θα κρατήσει τα επόμενους ε, μήνες ε, στο άμεσο μέλλον, διότι είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας, γιατί έχουμε πάρα πολλά αιτήματα που αφορούν αυτό το θέμα. Μη έχετε μήπως πρόθεση να, κάνε, να εισάγετε ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο για την ουδετερότητα. Ωραία. Λέει ο πρόεδρος θα απαντήσει σύντομα η κυρία Επίτροπος ε, τον πρώτο γύρο Ερωτήσα. Έχετε το λόγο. Πρώτη ερώτηση της κυρίας Τρότμαν. Ευρωπαίανα. Η είναι ένα πολύ σημαντικό, συμβολικό θα έλεγα πρόγραμμα δικό μας με εταιρική σχέση με τις κυβερνήσεις με τα πολιτιστικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, μουσεία, Μέχρι στιγμής είμαστε περίπου στα 8,5 εκατομμύρια αντικείμενα που υπάρχουν στο δίκτυο Ευρωπαϊάνα. Η συμβολή των κρατών μελών είναι άνηση. Κυρία Τρότμαν, ευχαριστώ τους Γάλλους, διότι τα μισά από τα αντικείμενα στην Ευρωπαϊάνα είναι γαλλικής προέλευσης. Λέω ευχαριστώ στους Γάλλους και λέω στους άλλους κουνηθείτε, κινηθείτε, δεν είναι φυσιολογικό. 50% της ευρωπαϊκής κουλτούρας δεν είναι γαλλική. Πρέπει και οι άλλοι να φροντίσουν έτσι ώστε η Ευρωπαία να είναι επιτυχία. Βέβαια, έχουμε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή δεν θα είναι πια ένα, απλώς ένα μωρό και θα αρχίσει να μπαίνει στην εφηβεία και θα συμβεί αυτό του χρόνου και τα επόμενα χρόνια φυσικά θα πρέπει τότε να αναζητήσουμε ε, εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Έτσι το Ευρωπαϊκό να γίνει αυτό που ανέκαθεν θέλαμε, ένας χώρος όπου ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία. Επιστημονικές εκδόσεις. Στις συζητήσεις για την ψηφιακή βιβλιοθήκη επί έτη φρόντισα να έχουμε επαφή με εμπειρογνώμονες σε πολλούς τομείς, πνευματικά δικαιώματα, τα ορφανά έργα όπως τα λέμε, επιστημονικές δημοσιεύσεις. Και οι εμπειρογνώμονες αυτοί με βόηθησαν ώστε να έχουμε, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα στην ιδιομορφία του κάθε τομέα. Γιατί τα μυθιστορήματα από μια μεριά, οι επιστημονικέ δημοσιεύσει ή τα παιδικά βιβλία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αν τα συγκρίνουμε, αυτό που μπορούμε να πούμε γενικά είναι οτιδήποτε ε, είναι ανήκει πια στον, στη δημόσια πρόσβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πρόσβασης Βέβαια αυτό είναι εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνουμε. Το κάνουμε ωστόσο. Και για τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί υπάρχουν όπως σας είπα ορφανά βιβλία που δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, υπάρχουν όμως και βιβλία που ε, των οποίων η, η, η έκδοση έχουν εξαντληθεί. Υπάρχουν δηλαδή τέσσερις, τέσσερις, τέσσερις ομάδες. Υπάρχουν τα βιβλία που ακόμα υπάρχουν στο εμπόριο. Εκεί πνευματικά δικαιώματα παίρνουν αμφισβήτηση στο εμπόριο. Μετά έχουμε βιβλία που ακόμα καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα αλλά έχουν εξαντληθεί. Δεν είναι διαθέσιμα. Είτε γιατί δεν μπορούν να γίνουν ψηφιακά, γιατί δεν γνωρίζουμε το συγγραφέα. Αυτά είναι τα ορφανά βιβλία πρέπει να υπάρξει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ορφανά αυτά βιβλία, γιατί είναι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινή κληρονομιάς μας που δεν μπορεί να περάσει στο ψηφιακό χώρο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν την δική μας ευρωπαϊκή λύση. Τρίτη ομάδα είναι τα out of print, τα εξαντλημένα, που καλύπτουν όμως ακόμα από πνευματικά δικαιώματα. Ε, εκεί είναι πιο εύκολο να βρεθεί η λύση. Και τέλος υπάρχουν όλα τα άλλα τα οποία ε, όπου δεν υπάρχουν πια πνευματικά δικαιώματα. Τέσσερις ομάδες λοιπόν. Και όταν είχαμε τη συζήτηση για τα Google Books είπα δεν χρειάζεται εδώ στην Ευρώπη να εφαρμόσουμε λύσεις άλλων υπήρων πρέπει να βρούμε δικές μας λύσεις. Ετοιμαζόμαστε εδώ και δύο χρόνια με όλους τους ενδιαφερόμενους ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τις δυνατές λύσεις. Το νέο Κοινοβούλιο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο ας φροντίσουν να υπάρξουν αυτές οι συγκεκριμένες λύσεις. Τώρα, προδιαγραφές και πρότυπα. Ως Ευρωπαίοι δεν τα πάμε και πολύ καλά όσον αφορά προδιαγραφές και πρότυπα. We could do better. Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιδόσεις. Έτσι ώστε κάποιος για να γνωθεί κάτι στην Ευρώπη οι δυσκολίες είναι πολύ πιο μεγάλες από ό,τι σε άλλες επίρρους. Γι' αυτό έχουμε την λευκή βίβλο, white paper, που αυτή τη στιγμή συζητιέται και πρέπει εμείς, και όταν λέω εμείς, ενώ το λέω επίτηδε, γιατί υπάρχουν πολλοί επίτροποι που ασχολούνται με το θέμα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πολλές πολιτικές. Μία πολιτική πρέπει να έχουμε, μία κοινή πολιτική ευρωπαϊκή που να εξυπηρετεί και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον τη βιομηχανία γενικότερα, όλο τον κλάδο, ιδιαίτερα όσον αφορά το, ε, το το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες. Πρέπει να, έχ, να υπάρχουν αποκλειστικά κονσόρσια και task force δυνάμεις, ειδικέ ομάδες μελέτης και δράσης όπως υπάρχουν αλλού. Φαντάζομαι ότι απάντησα κατά κάποιο τρόπο στο θέμα του περιεχομένου στο διαδίκτυο και των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι η συζήτηση που θα κάνουμε ειδικά για τα βιβλία είναι παρόμοια με τη συζήτηση με το άλλο είδους περιεχόμενο που διακινείται. Από τη στιγμή που θα υπάρχει η τεχνολογία, ε, η δομή θα είναι η ίδια. Η διαφοροποίηση λοιπόν που είχαμε στον αναλογικό κόσμο θα μετράει όλο και λιγότερο. Θα έχουμε δηλαδή συγκεκριμένες λύσεις για τον ψηφιακό κόσμο. Και σας είπα ότι η δουλειά αυτή δεν αρχίζει από το μηδέν. Ήδη είμαστε στη φάση εφαρμογής. Cloud computing. Αυτό όντως είναι κάτι το καινούριο και έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής όπως ήθεστε στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό για να βρούμε λύση γιατί αν δεν υπάρξει λύση προστασίας στο cloud computing γιατί εγώ θεωρώ ότι το cloud computing είναι ένα πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν θέλουν να επενδύσουν πάρα πολύ γιατί είναι μικρές. Θέλουν να τις κάνουν με το τρέχον σύστημα. Το cloud computing μπορεί να τους βοηθήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λύσει το πρόβλημα προστασία. Η δουλειά αυτή έχει ξεκινήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί και υπολογίζει στη βοήθειά σας. Η ουδετερότητα του δικτύου Δώστε μου λίγο παραπάνω χρόνο γι' αυτό. Διότι κυκλοφορεί το θέμα αυτό εδώ και κάμποσο καιρό. Από τότε που συζητήσαμε το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά δεν ασχοληθήκαμε ποτέ σοβαρά με αυτό, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόβλημα Πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά αμερικάνικο, διότι οι Αμερικάνοι έχουν ένα σύστημα υποδομής τηλεπικοινωνιών εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. είναι εντελώς απορριθμισμένο νομικά, δηλαδή δεν υπάρχει νομική νομικοί περιορισμοί με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις και πολύ μικρός ανταγωνισμός στην αγορά, στην Αμερική, που σημαίνει ότι ο πολίτης δεν έχει επιλογή του ESP, έχει αυτό που του προσφέρεται και τίποτα άλλο. Οι μεγάλες αυτές ομάδες λοιπόν έχουν εξουσία σε σχέση με το τι θα προσφέρουν ή τι δεν θα προσφέρουν στον πολίτη. Εμείς όμως στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια Έχουμε μια πολιτική τηλεπικοινωνιών ανοίγματος των αγορών. Υπάρχει ανταγωνισμός και ο καταναλωτής έχει επιλογή. Εδώ και χρόνια στην Ευρώπη έχουμε μια πολιτική που δίνει τη δυνατότητα στον εθνικό ρυθμιστή και στον ευρωπαϊκό ρυθμιστή, την Κομισιόν, να παίρνει μέτρα αν κάτι δεν πάει καλά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Μέχρι τώρα κανένας δεν έχει πάρει μέτρα. Επιπλέον, στο νέο πλαίσιο τηλεπικοινωνίες, δίνουμε μεγαλύτερη δυνατότητα στον εθνικό αριθμιστή να παρέμβει αν υπάρξει πρόβλημα. Οι Αμερικάνοι το είδαν αυτό και άρχισαν και αυτοί να κινούνται γιατί αυτό έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Προσέξτε λοιπόν. Όχι επειδή συζητάνε στην Αμερική το θέμα αυτό, μη θεωρούμε ότι το θέμα αυτό και το πρόβλημα αυτό είναι το ίδιο και για την Ευρώπη. Ευτυχώς δεν είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διότι σας θυμίζω κάτι που ανέκαθεν λέω ότι είναι απαράδεκτο οι ESP, οι πάροχοι αυτοί να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πόσες φορές ε, διαμαρτυρήθηκα όταν το Skype τον μπλοκάρισαν από πρόσβαση στο δίκτυο. Αυτό δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να έχουμε ένα διαδίκτυο ανοιχτό και θα το κάνουμε αυτό. Όπως βλέπετε κύριε Πρόεδρε, θα τη συζητήσουμε την ιστορία αυτή, αλλά για όνομα του Θεού δεν υπάρχει λόγος να εκνευριζόμαστε υπερβολικά. Αν εκνευρίζονται σε κάποια άλλη ήπειρο, άλλη ιστορία αυτή. Εμείς να λύσουμε το πρόβλημά μας στην Ευρώπη ως Ευρωπαίοι. Μην χρησιμοποιούμε τα σλόγγαν και τα συνθήματα των άλλων. ambient assistant living. Δύο ευρωβουλευτές έθεσαν το ερώτημα. Είναι αυτό ένα σημαντικό εργαλείο για να λύσουμε ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε που είναι η γύρανση του πληθυσμού. Όχι να το λύσουμε, να διευκολύνουμε τους ε, Η αντίδραση των κρατών μελών ήταν θετική επέβησαν περισσότερο από ό,τι είχαν πει αρχικά 600 εκατομμύρια ευρώ αν έχουμε περισσότερα λεφτά τόσο το καλύτερο αλλά δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά διότι πολλοί από αυτούς που ασκούν που εφαρμόζουν μάλλον τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ένας εύκολος τρόπος μερικές φορές τους βοηθάει παρά να, τους, να έχουν περισσότερα χρήματα. Αν το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι, μπορεί, ότι μπορούμε να είμαστε πιο ενεργοί στο μέτωπο αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε και θα έπρεπε και να αυξήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια εγώ συμφωνώ να το κάνουμε αυτό γιατί είναι ένα θέμα πάρα πάρα πολύ σημαντικό προστασία των δεδομένων, data protection. Ακόμα ένα θέμα που θεωρώ ότι θα σας ε, απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμη. Ξέρετε ότι στην Κομισιόν ξεκινήσαμε μια ανοιχτή διαβούλευση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πληροφοριών αυτό ξεκίνησε στις 9 Ιουλίου και θα συνεχιστεί αυτή η διαβούλευση μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Θα έχουμε πολύ αυστηρή νομοθετική ρύθμιση, θα έχουμε οδηγία ή θα το λύσουμε με ένα πιο ήπιο τρόπο. Αυτή η απόφαση δεν έχει λυθεί ακόμη. Ο επόμενος επίτροπος θα πρέπει να το συζητήσει αυτό με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Γιατί άλλο πράγμα <clears throat> με οδηγία και άλλο πράγμα ο κανονισμός. Με τον κανονισμό τα πράγματα γίνονται πιο γρήγορα. Για η οδηγία για να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες μέλη μερικές φορές χρειάζεται και πέντε χρόνια. Εδώ έχει σημασία η διάσταση χρόνος στην εφαρμογή των κανόνων. Οι εξελίξεις εδώ είναι πάρα πολύ γρήγορες. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Στο πακέτο Telecom έχουμε αυτή την υποχρεωτική κοινοποίηση των παραβάσεων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα άρθρο 4. Έχουμε ενισχυμένη προστασία όσον αφορά τα malware, spyware και τα cookies. Έχουμε νέα νομικά μέτρα κατά των spammers, αυτών που στέλνουν ε, χωρίς λόγο διάφορα email και την ε, διευκόλυνση στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του νέου άρθρου 15α. Όλα αυτά μας βοηθάνε να προστατεύουμε την ατομική σφαίρα, τη σφαίρα του ιδιωτική ζωής. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα τηλεπικοινωνιών, είναι γενικότερο θέμα. Βλέπετε, παραδείγματο χάρη, πόσο έντονα παρενέβην όταν είχαμε παραβάσεις σε συγκεκριμένες μορφές διαφήμισης, όπως θα έπρεπε να γίνονται ή να μην γίνονται. Στοχευμένη διαφήμιση. Targeted advertised. Εδώ έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες που λένε ο πολίτης θα πρέπει να έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων. Να γνωρίζει όμως τα δικαιώματά του. Πρέπει ο πολίτης δηλαδή να γνωρίζει τα δικαιώματά του και δεύτερον να εφαρμόζεται τα δικαιώματά του αυτού πρακτικά. Ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα με την Βρετανική κυβέρνηση έχουν πάει σε δικαστήριο για το περίφημο form, form system όπως το λένε. Δεν, με, πήγαμε σε δικαστήριο κατά του φόρμα, αλλά ως προς το πώς η Βρετανική κυβέρνηση εφαρμόζει τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας. Ε, με ε, έγκυρο χαρακτήρα, trusted sources. Η κατά νου έχουμε περισσότερο το σύστημα του κανονισμού. Όπως θα θυμόσαστε όταν αποκινούμε την Επίτροπο Κουνέβα ξεκινήσαμε τις κατευθύνσεις γραμμές της Ένωσης 5 Μαΐου, ένα από τα στοιχεία ήταν αυτό το θέμα των trusted sources, των έγκυρων πηγών. Τώρα αυτό ρυθμίζει, ε, μπορεί να λυθεί με αυτορύθμιση ή όχι. Προσωπικά, αν κάτι μπορεί να λυθεί χωρίς υπερβολική νομοθεσία, το προτιμώ. Αν μπορεί να ε, λυθεί με αυτορύθμιση, το προτιμώ. Αν όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε, οπότε θα πρέπει να το συζητήσουμε από κοινού, κύριε Πρόεδρε, διότι ε, πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνιστόσα. Πρωτοβουλία Ευρυζωνική, Broadband Initiative. Είμαι και χαρούμενη και στενοχωρημένη ταυτόχρονα. Χαίρομαι διότι όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε τα της ευρεία ζώνης και την πολιτική του φάσματος γενικότερα, πολλές κυβερνήσεις είπαν ότι δεν είναι πρόβλημα φάσματος ούτε ευρυζωνικό. Τώρα νομίζω όλοι συμφωνούν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Αν το 30% του πληθυσμού δεν καλύπτεται έχουμε πρόβλημα. Χαίρομαι λοιπόν για το ότι ε, ανέβηκε το επίπεδο συνειδητοποίηση. Αυτό όμως που δεν καταφέραμε ακόμα είναι να περάσουμε από τη συνειδητοποίηση στην πολιτική επένδυση. Και είμαι απογοητευμένη, διότι οι κυβερνήσεις που θα μπορούσαν να είχαν υποφεληθεί από το ένα δις που δώσαμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για την ευρυζωνική σύνδεση, ε, λοιπόν, πολλές κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα. Δηλαδή ακόμα στα προγράμματα δράσης δεν προβλέπουν την ανάγκη η ευρυζωνική λύση να βοηθήσει τις χώρες τους να βγουν από την κρίση. Και έχετε δίκιο. Όταν θα ορίσουμε τη νέα περιφερειακή πολιτική, η ευρυζωνική πρόταση καλύπτεται βέβαια από τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής. Εκεί θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές συνιστώσεις της πρότασης. Η αλλαγή, η ευρυζωνική αλλαγή. Broadband switch over. Γιατί επιμένω να περάσουμε πιο γρήγορα από τα αναλογικά στα ψηφιακά. Διότι χρειαζόμαστε αυτές τις συχνότητες για να έχουμε την ευρυζωνική ανάπτυξη και γι' αυτό η Κομισιόν θα κάνει αυτή την ανακοίνωση για το ψηφιακό μέρισμα στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται. Θα είναι ένα από τα τελευταία συγκεκριμένα μέτρα της σημερινής Κομισιόν. Έχει συμβολική σημασία λοιπόν. Το τελευταίο σημαντικό πράγμα που θα κάνει αυτή εδώ η Κομισιόν είναι το ψηφιακό, η ανακοίνωση για το ψηφιακό μέρισμα. Και χρειάζεται καλή προετοιμασία για την διάσκεψη για το φάσμα Μετά τη διάσκεψη οι κυβερνήσεις θα καταλάβουν ότι το φάσμα δεν είναι κάτι μικρό ότι το φάσμα, το σπέκτρουμ αφορά όλο, όλη την γεωγραφική επικράτεια της Ένωσης και συμφωνώ με αυτό που είπατε να ορίσουμε έναν οδικό χάρτη κατά κάποιο τρόπο ένα χάρτη, φύλλο, χάρτη πορείας όσον αφορά το ψηφιακό μέρισμα και το φάσμα τη διάσκεψη για το φάσμα Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Ντερκαστήγιο. Αν φέρουμε την ευρυζωνική πρόσβαση στους ηλικιωμένους ή σε περιοχές που σήμερα δεν καλύπτονται, αν δεν έχουμε περιεχόμενο και υπηρεσίες, τι ο λόγος. Και αν δεν έχουμε χρήστες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν, τί; είναι κυρίως ευθύνη των κυβερνήσεων. Να υπάρξει μια γνώση στη χρήση της ψηφιακής μεθόδου. Να καταπολεμηθεί δηλαδή ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Έρευνα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την έρευνα του ICT της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. 600 εκατομμύρια έχουμε στο τραπέζι μας για την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων, αλλά έχουμε και την ε, πρωτοβουλ... τις πρωτοβουλίες ε, κοινή ε, τεχνολογίας, τα JTIs, και σας διαβεβαιώ ότι κάθε παίκτη σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίξει το ρόλο του. Η Κομισιόν παίζει το δικό της, ο, ο τομέας της ε, βιομηχανίας το δικό του και αυτοί που δεν παίζουν το ρόλο του έτσι όπω θα έπρεπε είναι δυστυχώς τα κράτη-μέλη. Γιατί ε, πρέπει να το αναλύσω αυτό το γεγονός. Θα επανέλθω και το μόνο που μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω είναι να σας εκθέσω τα στοιχεία. Τα πράγματα, εκεί όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Και πρέπει τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι το, το, το πρόβλημα αυτό της, ε, της ανταποδοτικότητας είναι παλαιομοδίτικο. Δηλαδή ό,τι βάζω το παίρνω, διότι αυτή τη στιγμή αν βάλουμε σε ένα σύστημα ή αν δώσουμε, αν προσφέρουμε κάτι, το όφελος που έχουμε είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάζω μέσα ένα, δηλαδή προσφέρω ένα βιβλίο και παίρνω χι γνώση πίσω ας πούμε. Ε, εδώ από την, ε, το συντονισμό των πηγών και των προσφορών μας το όφελος για όλους θα είναι τεράστιο. Πριν από αρκετά χρόνια, την εποχή του πρόεδρου Κλίντον, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερικανική κυβέρνηση είχε αρχίσει να συζητάει την δυνατότητα να, να βγει το ICOM έξω από την επίβλεψη του, των Αμερικανών. προχωρούσαμε πολύ καλά, πολύ καλά, να βγει εκτός δηλαδή Αμερικανικού ελέγχου. Εν συνεχεία τον Νοέμβριο βγήκε ο Μπούς και όλα πάγωσαν. Όταν άλεξε η κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκέφτηκα ότι καλό θα είναι να προχωρήσουμε με αυτό το ζήτημα και το Μάιο. Στην ομιλία μου έκανα μία έκκληση στον πρόεδρο Ομπάμα να βγάλει το ICON εκτός αμερικανικής επίβλεψης. Να το βγάλει έξω από κάθε σύστημα επίβλεψης για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ελεύθερο ίντερνετ χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μετά από αυτό λοιπόν, το Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών υποστήριξαν support. Υποστήριξαν πλήρως αυτά τα οποία ζήτησε η Κομισιόν και η Τρόικα, οι δύο Προεδρίες και η Κομισιόν, το Σεπτέμβριο άρχισαν να τις διαβουλεύσεις, τις διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό σε μια-δύο μέρες και αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον oversight, επίβλεψη δηλαδή της αμερικανικής πλευράς επί του ICAM και ότι η Ένωση Πώς το λένε το GAG, μπορείτε να με βοηθήσετε, τι σημαίνει το GAG. Government και το κυβερνητικό, η κυβερνητική συμβουλευτική ομάδα Government Advisory Group, το λεγόμενο GAG, η κυβερνητική συμβουλευτική ομάδα Government Advisory Committee λοιπόν, Committee. Σα καλύπτει τέσσερις πλατφόρμες με εμπειρογνώμονες οι θα ονομάζονται από την Επιτροπή αυτή τη συμβουλευτική με διευθύνοντα σύμβουλο από την ICAM για να επιβλέπει ακριβώς αυτές τις ε, τέσσερις λειτουργικές πλατφόρμες. Η εξέλιξη αυτή, η νέα δομή θα έχει μεγάλη επίπτωση για μας το Κοινοβούλιο γιατί η συζήτηση που θα γίνει στο Sharm el θα έχουμε εμεί μεγαλύτερο κύρος, ο ρόλος μας θα είναι πιο σημαντικό γιατί θα πρέπει να, να γεφυρώσουμε το GAC αυτό, το GAC δηλαδή και την κοινωνία των πολιτών ώστε αυτό το νέο σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει διότι έχουμε το νέο αυτό σύστημα θα το έχουμε δηλαδή μπροστά μας σε χαρτί και θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε δράση είναι λοιπόν μια ιστορική στιγμή αυτή για την κοινότητα του διαδικτύου και είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε την δυνατότητα με τους Αμερικανούς να συμβαδίσουμε και με άλλα μέρη του κόσμου που πιστεύουν στην, στο ελεύθερο διαδίκτυο και πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χέρι με χέρι στη δημιουργία των θεσμών για να λειτουργήσει αυτό το ελεύθερο ίντερνετ. Είδατε μερικές φορές αν, αν πραγματικά ε, το επιδιώξεις, πατήσεις το πόδι δηλαδή, έχουμε επιτυχίες μεγάλες. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Τώρα, βλέποντας το ρολόι μας εδώ και τον κατάλογο των ομιλητών, σας παρακαλώ να είμαστε σύντομοι. Το πλεονέκτημα είναι ότι βεβαίως λαμβάνουμε πολύ λεπτομερείς πληροφορίες για τις εργασίες μας, αλλά παρακαλώ όχι, όχι, μακρηγορία, η κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικό με την ασφάλεια που είναι απαραίτητη στη κοινωνία της πληροφορία. Και εδώ αναφέρομαι σε καταναλωτές και σε παρόχους υπηρεσιών, providers δηλαδή. Μπορούμε να διαβάσουμε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 90% των ε, κοινοφελών υπηρεσιών, 90 παρέχουν οι υπηρεσίες και ηλεκτρονικά. Δυστυχώς όμως, όπως ισχύει και με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπογραφή, δεν έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργικότητα. Δεν είναι συμβατά τα συστήματα. Γνωρίζουμε ότι έχετε ορισμένες μελέτες που λέγουν ότι μέχρι το 2009, το τέλος του έτους, θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, και το 2010 τελικά να καταλήξουμε σε μια κοινή υπηρεσία για πιστοποίηση και έγκριση ηλεκτρονικής υπογραφής πανευρωπαϊκά. Πού βρίσκεστε τώρα σχετικά, τι ε, προγραμματίζετε ως ενέργειες για τους επόμενους μήνες και ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΝΙΣΑ εδώ, γιατί γνωρίζουμε ότι η εντολή λύγει τέλη του 2012 και υπάρχει ένα ζήτημα ασφαλείας όλο και πιο οξύ ε, στο ίντερνετ γιατί θα πρέπει οι ε, καταναλωτές να εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Γι' αυτό φοβάμαι, μάλλον εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος και η διάρκεια της ενίσα θα πρέπει να παραταθεί. για να αντιμετωπίζονται καλύτερα κάποια ζητήματα ασφαλείας ή όταν έχουμε επιθέσεις ε, στους υπολογιστές. Και είναι και θέμα υποδομών. Οι ηλεκτρονικές υποδομές και οι τηλεπικοινωνίες θεωρούνται ευαίσθητες. Ξέρω ότι υπάρχει οδηγία για τις υπηρεσίες που προβλέπει ότι από το 2010 ε, οποιαδήποτε εταιρεία θα έχει ωφέλη, θα μπορεί να υποφελείται μάλλον από την πρόσβαση σε δημόσια υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Τι σχεδιάζεται εκεί λοιπόν. Και μια τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αναθεωρήσει την οδηγία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright στην κοινωνία της πληροφορία. Γιατί το ρωτώ αυτό. Γιατί η σημερινή οδηγία έχει ερμηνευθεί διαφορετικά από χώρα σε χώρα και έχουμε νομολογία στα κράτη-μέλη σχετική που διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που το εκμεταλλεύονται και οι χρήστες δεν έχουν πάντα την ίδια πρόσβαση. Αλλά υπάρχει και η διασυνοριακή ε, πρόσβαση. σκέφτεστε αυτό να αναθεωρήσετε την οδηγία για το copyright στο δίδυκτο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρβάλιο. Δεν έχω. Ευχαριστώ. Ε, δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ερώτηση πρώτη. Μιλήσατε για τα κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες με συμμετοχή της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων. Με τα πανεπιστήμια τι γίνεται κύριε Ρέντινγκ. Εγώ ήξερα ότι βασικός στόχος ε, αυτών των πρωτοβουλειών είναι να προαχθεί η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή της βιομηχανίας. Εντάξει. Αλλά τι γίνεται με τη συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι στη βάση του τριγώνου της γνώσης και της καινοτομίας για την Ευρώπη. Γενικά γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες για τη συμμετοχή των πανεπιστημίων σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτές τις πρωτοβουλίες, ιδίως σε μικρές χώρες και μεσαίες χώρες. Ε, πώς έχει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα της κοινωνίας πληροφορίας για τις κοινέ ε, τεχνολογικές ε, προσπάθειες. Στη συνέχεια, Τι γίνεται με την ευρυζωνικότητα στα πλαίσια των σχεδίων ανάκαμψη οικονομία. οικονομίας. Ανησυχώ από αυτά που ακούω από την Επίτροπο. Μας είπατε ότι σας απογοήτευσε το γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσει δεν έχουν ακόμα αξιοποιήσει τα προγράμματα δράση του ή δεν τα έχουν ε, ολοκληρώσει και χάνουν χρήματα. Και αυτή η χρηματοδότηση αφορά το 2009 και 2010 θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για να δούμε τι γίνεται με αυτή τη χρηματοδότηση. Ποιος τη διαχειρίζεται. Σε κεντρικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες ή μήπως τα κράτη-μέλη ανάλογα, όπως τα διαρθωτικά ταμεία για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κολάς Καμποβίνσκα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα το, της, το, του της Ευρωζωνικής Σύνδεσης στο, στην Πολωνία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου όχι 30%, 70-80-90% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση. Τώρα το 2013 μπορεί να μας φαίνεται πάρα πολύ κοντά, αλλά για αυτούς φαίνεται, τους ανθρώπους είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτό το θέμα συντονισμένα, διότι καλύπτεται από πολλές επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Ε, είπατε ότι πρέπει και στα δικά μας τα κράτη να πιέσουμε για την ανάπτυξη του συστήματος. Ίσως λοιπόν οι ευρωβουλευτές μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από τη συζήτηση, να καταβάλουν περισσότερες δυνάμεις. Πρέπει να υιοθετήσουμε, να εγκρίνουμε και τον προπολογισμό του χρόνου τι μας προτείνει λοιπόν η Κομισιόν. Πέστε μας εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα της Κομισιόν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μόνο θεσμικά μέσα, αλλά υπάρχουν και άτυπα ε, ήπια μέσα, παραδείγματο χάρη, το να ξεμπροστιάσουμε κάποιον φορέα ο οποίος ε, αδρανεί, ο οποίος δεν κάνει τίποτα για το θέμα αυτό. Ε, επίσης, έχουμε πάρα πολλά προγράμματα που ακροβατούν, που είναι θνησιγενοί διότι δεν έχουν αρκετή χρηματοδότηση. Αν λοιπόν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτά τα προγράμματα, ίσως μπορούμε να τα ξαναζωντανέψουμε. Ας, βάλουμε, ας καθίσουμε λοιπόν όλοι μαζί και σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο πρακτικά μέτρα. Εν συνεχεία, ουδετερότητα του ίντερνετ. Έχω λάβει αρκετές επιστολές σχετικές με αυτό το θέμα και εδώ πέρα θέλω να πω ότι κυρίαρχη θέση έχουν οι προμηθευτές θα ήθελα να σας εξέσω ορισμένα σχόλια τα οποία έλαβα από τους ψηφοφόρους οι οποίοι λένε ότι κυρίαρχοι προμηθευτές μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο και, και να επηρεάσουν την καινοτομία. Αυτό έχει σχέση και με το άρθρο 21 της Οδηγίας Σφαιρικών Υπηρεσιών ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Δεν θέλουμε λοιπόν οι κυρίαρχοι προμηθευτές ε, που έχουν δεσπόζουσα θέση να επέμβουν και στο περιεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, για αυτή την ε, πολύ περιεκτική παρουσίαση. Είσαστε μία από τις πιο αποτελεσματικές επιτρόπους ε, και το βλέπουμε αυτό από τις πολλές εμφανίσεις πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε αναλάβει. Μιλήσατε για την εξάλληψη των διαφορών μεταξύ των αστικών και υπεθρίων περιοχών και βελτίωση της πρόσβασης στην ύπεθρο. Δυστυχώ, πολλέ πρωτοβουλίε δεν προχωρούν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε παρόλο που υπάρχουν πιστώσει για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως ε, οφείλεται ε, στο ότι οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν καλυφθεί από το πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης και των συναφών πολιτικών. Δεν έχουν ενταχθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω σε, ένα, μια περίοδο κρίσης να προωθήσουμε αυτές τις, πρωτο, τις επενδύσεις. Ίσως ορισμένες χώρες δεν έχουν κατανοήσει ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ότι μέσω αυτού της, της ευρυζωνικής θα, μας, θα μπορέσουμε να διευκολυνθούμε στην έξοδό μας από την κρίση. Το συμφωνείτε με μένα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, ο κύριος Γκέμπαρντ έχει το λόγο. Ο κύριος Ανρί Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ για την ακρίβεια και την πυκνότητα της απάντησής σας. Θα ήθελα, μου επιτρέπετε, να επανέλθω στην προτεραιότητα που υπογραμμίσατε κι εσείς και είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σήμερα δεν έχουμε ένα μόνο χάσμα, είναι τριπλό το χάσμα. Μιλήσατε για το χάσμα ε, ανάμεσα στην Ήπεθρο και στις πόλεις και την κάλυψη της Ήπεθρου. Όντως δεν καλύπτεται το 30% των κατοίκων που ζουν εκεί και είναι και σκάνδαλο αλλά και βαριά οικονομική αναπηρία. Υπάρχει όμως και άλλο χάσμα, εξίσου σημαντικό για μένα, που είναι το ε, κοινωνικό χάσμα. Μιλήσατε για ε, ψηφιακό αναλφαβητισμό. Σήμερα στις πόλεις μας, στα αστικά μας κέντρα, έχουμε πραγματικά ένα χάσμα μεταξύ εκείνων που είναι πλούσιοι σε γνώση, σε πληροφορίες και εκείνων που είναι σε φτωχοί σε γνώση. Και αυτή η φτώχεια έρχεται ε, να προσθεθεί ε, ως επιπλέον αναπηρία σε πολλά άλλα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Ε, σας βέβαια αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων και το είπατε, αλλά δεν υπάρχει καμιά ειδική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και ένα τρίτο χάσμα που υπάρχει και αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό είναι διαφορά βορρά-νότου. Υπάρχει ανισότητα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και τις πιο φτωχές ανάμεσα στις αναδυόμενες αλλά και στις πλουσιότερες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορά βορανότου που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Εμείς που είμαστε η πρώτη οικονομική και εμπορική δύναμη στον κόσμο δεν μπορούμε να διαφορούμε για αυτό το χάσμα που επίσης ε, οικονομικά θα είναι επιβαρυντικό. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόγια ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, αναγνωρίζω ότι η ώρα έχει περάσει, θα είμαι τηλεγραφική. Θα ήθελα απλώς να πω στην κυρία Ρέντινγκ ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προβλήματα αυτά και θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιε σαφεί απαντήσεις. Συνήθω οι απαντήσεις είναι πολύ συγκεκριμένε στις ερωτήσεις μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Τρία σχόλια έχω μόνο. Ελπίζω η Κομισιόν να επιμείνει στο roaming. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του σώματος και που μας επιτρέπει να δείξουμε ακριβώς στους πολίτες μας ε, τι μπορούμε να κάνουμε Πιστεύω ότι η ενδιάμεση έκθεση και αναθεώρηση θα συνεχιστεί. Όσον αφορά το φάσμα, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Πιστεύω ότι μερικές χώρες, όπως και η δική μου, ε, ε, το απελευθερούμενο φάσμα ε, το κρατάνε μυστικό. Κρατούν αυτή την ευκαιρία μυστική. Δεν την αποκαλύπτουν Ίσως, ε, ναι, πραγματικά πιστεύω να υπάρξει μια συντονισμένη κοινοτική δράση, διότι πολλές χώρες έχουν αποκρύψει αυτή τη δυνατότητα. Ιδίω χώρες όπου το σύστημα πληροφορικής τους είναι, ε, δεν είναι ομαλό ε, προσπαθούν να αποσιωπήσουν αυτή τη δυνατότητα, διότι αυτό το απελευθερωμένο φάσμα θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και ε, πιο ευρείας πρόσβασης. Μην ξεχνάμε και τα δικαιώματα των πολιτών. Το αναφέρατε και είναι σημαντικό. Ή τα δικαιώματα των καταναλωτών μας. Δεν είναι μόνο ο έλεγχος των διαφημίσεων ή των δεδομένων, η προστασία, η ιδιωτική φύση των δεδομένων. Όλα αυτά αποτελούν μια γκρίζα, ένα γκρίζο τομέα, γκρίζα περιοχή, συγκεχημένη, μπερδεμένη και γίνονται πάρα πολλές παρανοήσεις και παραπληροφόρηση υπάρχει επίσης σε αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια διατομεακή προσέγγιση, τηλεποκοινωνίες, πολίτες, καταναλωτές και αρμόδιοι φορείς. Υπάρχουν και πολλοί εμπορικοί πειρασμοί να εκμεταλλευτούν τις αμφιλεγόμενες, τους αμφιλεγόμενους τομείς. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν αυτό το θέμα και στο Ευχαριστώ. κυρία Ποδηματά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ και εσάς για την ε, περιεκτική σας εισήγηση και τις εμπεριστατωμένες ε, απαντήσεις σας. Είναι γεγονός και κατά τη δική μου άποψη ότι ο συνολικός απολογισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια είναι θετικός πέρα από επιμέρους παραλήψεις καθυστερήσεις και προβλήματα. Ε, δεν αναιρείται το γεγονός ότι έχουν υπάρξει όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ σημαντικά ωφέλη στους ευρωπαίους πολίτες είτε αυτό αφορά στον κανονισμό της περιαγωγής είτε αυτό αφορά στο, στο κόστος της σταθερής ή και της κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτως, ε, ανεξαρτήτως της περιαγωγής. Κυρία Επίτροπε, αναφερθήκατε στην ε, εισήγησή σας και στην επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες τα περίφημα ε, mss. είναι μια συζήτηση που την είχαμε πέρσι την άνοιξη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ήθελα να θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είχε υπογραμμίσει σε ό,τι αφορά στα κριτήρια επιλογής των φορέων δύο στοιχεία. το πρώτο ήταν η υποχρέωση των επιλεγμένων φορέων να παρέχουν ε, πανευρωπαϊκές υπηρεσίες και το δεύτερο να υπάρχει διασφάλιση ε, του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών σε περίπτωση ε, φυσικών καταστροφών. τον περασμένο μάιο επελέγησαν οι δύο φορείς για να αναλάβουν την παροχή κινητών δορυφορικών υπηρεσιών και πολύ σύντομα μετά την επιλογή του η μία από τις δύο εταιρείες ανακοίνωσε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα κάποιες δυσλειτουργίες ε, στο δορυφόρο. ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με δεδομένο ότι αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν βασικό στόχο όχι μόνο της, ε, της κοινωνίας της πληροφορίας για μια εξελιγμένη γενιά υπηρεσιών αλλά όπως είπα και πριν συνδέονται άμεσα και με τις ε, υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών εκεί δηλαδή που τα επίγεια ε, μέσα επικοινωνίας είτε δυσλειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου και έχω στο μυαλό μου τις ε, πρόσφατες και δυστυχώς επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό νότο κυρίως τα καλοκαίρια με τις, ε, με τις δασικές πυρκαγιές. ήθελα λοιπόν κύριε επίτροπε να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν ε, στο ζήτημα αυτό. Έχουν αρθεί τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν. Υπάρχει πιθανότητα η Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ε, απονομή των ε, αδειών για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στους υποψηφίους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Μπαλσίτης. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι έχετε επιτύχει Έχετε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στους τομείς σας, το ίντερνετ, ευρυζωνική σύνδεση, ε, ασφάλεια οδική ε, και και οικονομικές επιτυχίες βεβαίως ε, αλλά και έχετε σώσει με τα, μέτρα αυτά πολλές ζωές. Αυτή τη στιγμή βέβαια βρισκόμαστε μέσα σε μια οικονομική κρίση και σήμερα κάθε κυβέρνηση μπορεί να λάβει τις αποφάσεις της αν θέλει ή όχι να συνεχίσει ορισμένα προγράμματα αλλά στο μέλλον αυτή η ελευθερία στη λήψη των αποφάσεων πρέπει να παρακολουθείτε με προσοχή διότι αντιμετωπίζουμε ε, μία, έναν πολύ ανταγωνιστικό κόσμο και πρέπει να προβάλλουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες αποφάσεις πρέπει να τις πάρουμε όλοι μαζί από κοινού. Ιδίως ε, στον τομέα των ε, της ε, τεχνολογίας της πληροφορικής πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν συνεχίσει τις προσπάθειές τους συνήθως επειδή λείπουν τα χρήματα. Ίσως λοιπόν η Κομισιόν θα πρέπει να παίξει έναν πιο επικοδομητικό ρόλο ε, αναλογιζόμενοι όχι μόνο τα μελλοντικά ωφέλη αλλά και τις ζημίες που μπορούν να ληφθούν από ορισμένε αποφάσεις σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι για αυτή τη δέσμη των ερωτήσεων και καταλήγοντας θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πίτωπο να απαντήσει στον τελευταίο γύρο. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, διότι πολλές ερωτήσεις ή τμήματα ερωτήσεων ε, έχουν ήδη απαντηθεί από μένα προηγουμένως. Όσον αφορά την ασφάλεια, η ΕΝΙΖΑ έχει λάβει την ε, εντολή της, δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί τα τρία θεσμικά όργανα αν υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε περαιτέρω την εντολή αυτή ή όχι. Δεύτερο ερώτημα που αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή που πάει άπτεται της ασφάλειας, έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται κυρίως στη διαλειτουργικότητα, διότι ξέρετε ότι τα βασικά δικαιώματα καλύπτονται στο πλαίσιο της επικουρικότητας και πρέπει να σεβαστούμε την, επικουρικότητα, την αρχή της επικουρικότητας στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τα GTIs και τα πανεπιστήμια, Α, όχι, ε, το copyright λέει, διορθώνεται κύριε Επίτροπο. Η εθνική νομολογία διαφέρει από κράτη σε κράτη. Γι' αυτό ακριβώς ε, εκδώσαμε μία πράσινη βίβλο. Α, θα εκδώσουμε μία πράσινη βίβλο, ο, κύριος, ε, ο Επίτροπος κύριος Μαγκρίντι και εγώ, και στην πράσινη αυτή βίβλο θα αναφέρουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, ένα follow-up δηλαδή, και για να εδραιώσουμε μία σιγουριά και μία ασφάλεια σε όλα αυτά τα συστήματα και ένα ακλόνητο, ένα σταθερό σύστημα παροχής αδειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καυτό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε τους επόμενους μήνες. GTIs τώρα και πανεπιστήμια. Η έρευνα της τεχνολογίας, τεχνολογική έρευνα μάλλον, είναι, πολύ, είναι θεμελιώδης και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος χρηματοδοτείται από τον τομέα, από τον ε, βιομηχανικό τομέα, διότι χρησιμοποιεί τις δικές του πηγές. Τα πανεπιστήμια και τα, εργαστήρια μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, έρευνες οι οποίες γίνονται συντονισμένα από διάφορους αρμόδιους φορείς και η χρηματοδότηση προέρχεται από το GTI, από το GTI για να χρηματοδοτήσουν τους φορείς που δεν έχουν αρκετά δικά τους, δικές τους πιστώσεις και έτσι μπορούν να ε, διοχετευτούν περαιτέρω στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η διαδικασία. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου ή την υποβοήθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου με προηγμένα συστήματα. Σας είπα ότι κατά μέσο όρο 30% των κατοίκων της υπέθου δεν καλύπτονται ευρυζωνικά. Δεν λέω ότι σε ορισμένε περιοχέ σαφώ είναι πολύ υψηλότερα τα ποσοστά, αλλά στο πανευρωπαϊκά είναι γύρω στο 30%. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να πατήσουμε το πόδι μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το ένα δις ε, που, ε, το οποίο έχουμε ζητήσει αυξάνεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αν λάβουμε υπόψη όλη τη χρηματοδότηση του, της υπαίθρου. Βεβαίως αυτά δεν φτάνουν. Το καταλαβαίνω αυτό όταν μιλάμε για 30% μόνο ευρυζωνική κάλυψη. Το 70% χρειάζεται πολύ περισσότερες πιστώσεις. Γι' αυτό πρέπει και τα κράτη-μέλη να πιέσουν το, τους τομείς τους, τους αρμόδιους τομείς, βιομηχανίας, οικονομίες, ή να προσφέρουν και κρατικές ενισχύσεις για να μπορέσουν να προχωρήσει αυτά τα προγράμματα. Τώρα το ένα δις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, νομίζω ότι οι Υπουργοί Γεωργίας πρέπει να καταλάβουν επιτέλους τα ωφέλη ε, της ε, διάχυσης του ευρωζωνικού συστήματος στις υπαίθριες, ε, στην περιφέρεια. Θα αναπτυχθεί η πεθρός αλλά και οι επιχειρήσεις, η παραγωγή, εκμεταλλεύσεις, όλοι θα ωφεληθούν στην ύπεθρο από το ευρυζωνικό, την ευρυζωνική πρόσβαση. Πιστεύω ότι ανα, απάντησα ήδη στο θέμα της ουδετερότητας του δικτύου και την πρόταση να συνεχίσουμε στο μέλλον όπως κάναμε και στο παρελθόν με τη μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Να συνεργαστούμε έτσι ώστε τα συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν στην Ευρώπη να μπορούν να αντιμετωπιστούν με σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένες λύσεις. Το ζήτημα της ε, ηλεκτρονικής πρόσβασης ή accessibility. Στις 5 ε, Μαΐου μαζί με την ε, κυρία Κούνεβα συζητήσαμε το θέμα αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει να, συζητήσουμε την νομοθετική πράξη ηλεκτρονικής πρόσβασης έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα πρότυπά μας σε αυτά των Αμερικανών για να βελτιώσουμε και τη δική μας λειτουργικότητα. Λοιπόν, προσαρμογή των προτύπων με τα αμερικανικά. Τώρα, το χάσμα πάλι το ευρυζωνικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάσμα μπορεί να το κάνουμε με πιλωτικά προγράμματα αλλά πρέπει να γίνει αυτό οριζοντίως η αντιμετώπιση μας υπάρχει χάσμα ε, όσον αφορά τον αλφαβητισμό την, τον ψηφιακό αλφαβητισμό ακόμα και αν έχουμε μια γενική κάλυψη ευρυζωνική η απορρόφηση είναι μόνο 50%. Γιατί? Υπάρχει το θέμα του περιεχομένου πολλές φορές, το πρόβλημα του περιεχομένου, της διαλειτουργικότητας και των υπηρεσιών. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε το, την αναλογία κόστους-οφέλους, πρέπει τα, τα online contacts να γίνουν πιο εύκολα και να αυξήσουμε τον ψηφιακό αλφαβητισμό. Τώρα, όσον αφορά το χάσμα βορρά-νότου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε το ε, Internet Government Forum, ένα κυβερνητικό φόρουμ στο διαδίκτυο για να εξετάσει το πρόβλημα της ανάπτυξης σε άλλους υπήρους. Εγώ προσωπικά κατέβαλα μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη του, της ευρυζωνικής ε, πρόσβασης στην Αφρική. Προχωρούμε καλά, αλλά χρειαζόμαστε μια δυνατή, δυνατές κυβερνήσεις, ε, υπουργούς, ε, αποφασισμένους υπουργούς τηλεπικοινωνιών που θέλουν να προχωρήσουν τα συστήματα αυτά έτσι ώστε η Ευρυζωνική Σύνδεση να καλύψει όλους τους πολίτες. Ε, Και κοιτάζω προς την κυρία Τράουτμαντ, η οποία είναι πρωταγωνίστρια ε, στα θέματα αυτά στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί πάλι μια ισχυρή ομάδα ευρωβουλευτών ε, που θα ηγηθούν της ευρωπαϊκής προσπάθειας στο Σάρμελ el οι συχνότητες οι συχνότητες, το θέμα των συχνοτήτων πρέπει να συντονιστεί και γι' αυτό ε, βασίζομαι στην διάσκεψη για τις συχνότητες ε, που θα οργανώσουμε με το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι θα προκύψει ένα επικοδομητικό αποτέλεσμα. Για όλες, αυτά, αυτό ισχύει για όλες τις πολιτικές μας. Ο καταναλωτής, ο τελικός χρήστης, ο τελικά ωφελούμενος είναι πολύ, ε, ε, έχει πάντοτε πολύ ε, προταρχική πρωταρχική θέση στην ατζέντα μας και προς αυτούς προσβλέπουμε πάντοτε. Μία άλλη επιτυχής ε, προσπάθεια ήταν ε, οι κινητές ε, υπηρεσίες, οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, το MM, MSS, Mobile Satellite Services. Στις 13 Μαΐου υιοθετήθηκε η απόφαση και έχουμε 24 μήνες περιθώριο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος. Ε, θα παρακολουθήσουμε λοιπόν την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και την χρήση των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των διαφόρων κρατών μελών. Το σύστημα MSS λοιπόν. Η τελευταία ερώτηση τώρα. Συμφωνώ απολύτως. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να επανέλθουμε στον παλαιομοδίτικο εθνικισμό. Πιστεύω, όλοι τον έχουμε ξεπεράσει. Ε, πιστεύω ότι πολλές χώρες ε, δεν έχουν βγει ακόμα από την κρίση. αλλά άλλες χώρες που, ε, που βγαίνουν από την κρίση με, τις, με το μίνιμουμ των ζημιών δεν θα μπορούσαν να το είχαν επιτύχει αν δεν είχαν την ευρωπαϊκή Ελληλεγγύη να, τους, να τις υποστηρίξει. Ε, δείχνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ελληλεγγύη ακριβώς τι, μπορεί να, τι θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει, τι μπορεί η Ευρώπη να καταφέρει όταν είναι αποφασισμένη και θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα και σχόλια και ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για τις εμπεριστοκομμένες στις απαντήσεις πολύ χρόνο διέθεσε για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και πιστεύω ότι πολύ καλά κάναμε διότι με αυτή την ε, εντελεχή συζήτηση ε, καταφέραμε να συζητήσουμε πολλές ε, πτυχές του ζητήματος σε βάθος. Τώρα έχουμε το, τη διακοπή μας, θα συναντηθούμε το απόγευμα, όλοι χαρούμενοι.